σας καλωσορίζω στη δεύτερη αυτή δημόσια συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ που συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Γεωργίας και τον Πρόεδρό της κύριο Ντεκάστρο και τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Γεωργία κύριο Τσόλο. Και τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 12 Οκτωβρίου η Κομισιόν παρουσίασε μία δέσμη μέτρων για το μέλλον της ΚΑΠ για τη μεταρρύθμιση αυτής και τον Οκτώβριο επίσης έγινε συνεδρίαση του Συμβουλίου σε πρώτη της ανάγνωση το 10 Νοέμβριο συζήτηση για τις άμεσες πληρωμές και θα επαναληφθεί αυτή το Δεκέμβριο όπου θα συζητηθεί και το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ταυτόχρονα κατά την άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών στο Βρόθουα αποφασίσαμε να οργανώσουμε ανοιχτές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την, το μέλλον της ΚΑΠΗ. Η πρώτη τέτοια συζήτηση έγινε στις 7 Νοεμβρίου με συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας από ενωσιακές χώρες και εθνικούς βουλευτάς. Σήμερα Επίσης έχουν προσέλθει οργανώσεις γεωργών και εδώ ο κύριος Ντεκάστρο έχει κάνει μια πρόταση. Μου είπε ότι δεν έχουν, έρθει, δεν έχουν προσκληθεί όλες οι αγροτικές οργανώσεις αγροτών στην Ευρώπη, αλλά εμείς προσκαλέσαμε πάνω από 50 ούτως ή άλλως. Όχι μόνο τους εμπορευομένους γεωργικά προϊόντα αλλά και παραγωγούς. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να προσέλθουν όλοι ή να προσκληθούν όλοι οι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων. Αν λοιπόν κάποιον δεν βλέπετε, ίσως είναι γιατί δεν θεωρεί ότι ο ίδιος ότι τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα που συζητάμε. Στις 19 Δεκεμβρίου θα γίνει η τρίτη τέτοια συζήτηση χάρη στον κύριο Ντεκάστρο και κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο, τη Σύνοδο, θα γίνει και η σύνοψη τον Ιανουάριο. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας. Τώρα σε λίγο θα δώσω το λόγο στον κύριο Συμπρόεδρο Ντεκάστρο που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και μετά στον κύριο Επίτροπο. Και μετά θα μιλήσουν οι εισηγητές και οι συγγήτριες. Ύστερα δε έχουν γραφεί 25 ομιλητές και ομιλήτριες που θα έχουν 4 λεπτά έκαστος και εκάστη. Ελπίζω ότι μέχρι τις 6 θα τελειώσουμε. Αν περισσεύει χρόνος θα κάνουμε και οφθαλμοθυρία Catch the Eye. Πάντως μέχρι τις 6 πρέπει να έχουμε τελειώσει τη συζήτηση. Και να βγουν τα συμπεράσματα. Τώρα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ντεκάστρο. Ευχαριστώ αγαπητέ Μάρεκ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχουμε την ευκαιρία συμμετοχής ε, του αγροτικού κόσμου, από τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις, τις μη κυβερνητικέ και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μάρεκ Σαβίνσκι, ο οποίος οργάνωσε αυτή την ημερίδα έτσι ώστε να λάβουν το λόγο όλες οι οργανώσεις. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον Επίτροπο Τσόλος, ο οποίος είναι έτοιμος να προωθήσει έναν επικοδομητικό διάλογο. Πριν αρχίσει το νομοθετικό έργο, θέλουμε να ακούσουμε την κοινωνία των πολιτών, τις αγροτικές οργανώσεις, τα διάφορα θεσμικά όργανα και φορείς που θα συναποφασίσουν την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που αφορά μία εντελώς διαφορετική πορεία. Υπάρχει και το θέμα της διατροφικής ασφάλειας και των ελλείψεων στην αγορά. Υπάρχει μεγάλος κλειδονισμός των αγορών που μπορεί να γίνει ένα συστηματικό φαινόμενο. Η διατροφική προμήθεια είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και οι αγρότες χρειάζονται νέα μέσα έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μία έκρηθμη κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στις προμήθειες και επίσης να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να δούμε θέματα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που μας απασχολούν αυτά τα χρόνια. Χρειαζόμαστε όμως μία βιώσιμο, βιώσιμη γεωργία από οικονομικής πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα φέρουμε ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, έτσι ώστε να προσφέρουμε στους αγρότες μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυτή πρόκληση. Να παράγουν περισσότερο, μολύνοντας λιγότερο. Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νέα ΚΑΠ, έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο δυνατή οι αγρότες και παράλληλα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αγορές οι οποίες έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω ζημίες. Όπως ήδη υπογραμμίστηκε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούμε μια φιλόδοξη πορεία με δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας από τον George Lyon και από έναν άλλον εισηγητή. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή των πολιτών και μαζί με το Συμβούλιο θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την νομοθετική οδομαβάση αυτές τις δύο εκθέσεις, Lion και Des. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, η Ολομέλεια ενέκρινε τις δύο εκθέσεις που προανέφερα. Στις πρώτες συζητήσεις που έγιναν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου, την οποία προεδρεύω, θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθήσει την παραγωγή έτσι ώστε να επικαιροποιήσει τα δεδομένα με βάση τις αλλαγές που επέρχονται έτσι ώστε η ΚΑΠ να είναι πιο ευέλικτη στο μέλλον για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των αγορών που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θα ζητήσουμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση μια συμφωνία η οποία θα ε, γίνει το συντομότερο δυνατόν. Η σημερινή πρωτοβουλία, είμαι πεπισμένος αγαπητέ Μάρεκ, θα συνεισφέρει άμεσα με βάση την κοινή αυτή πορεία περισυλλογής μαζί με την κοινωνία των πολιτών και τον αγροτικό κόσμο. Αυτός ο ανοιχτός διάλογος θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε τα σημεία σύγκλησης για να μπορέσουμε να δώσουμε συνετές αποφάσεις με βάση τη συγκυρία που γνωρίζουμε. Έτσι η εργασία θα είναι σημαντική και χρήσιμη για τον αγροτικό κόσμο αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παόλο, για την εισαγωγή στο θέμα μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρικ. Και ευχαριστώ την Επιτροπή Γεωργίας που έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή τη διάσκεψη που ακολουθεί τη διάσκεψη που οργανώθηκε ήδη από την ε, ε, Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου και στις 19 19 Δεκεμβρίου ε, θα οργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διάσκεψη όπου θα είστε προσκεκλημένοι και θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των επιστημονικών ε, κλάδων για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλες τις προτάσεις και τις αναλύσεις για αυτό το θέμα. Θα κλείσουμε δηλαδή τις, ε, τον κύκλο των τριών συναντήσεων, τη σημερινή που οργανώνει το Συμβούλιο, την άλλη που έχει οργανώσει το Κοινοβούλιο και την επόμενη που θα οργανώσει η Επιτροπή. Πολύ σύντομα, θέλω να αναφερθώ στο περιεχόμενο των προτάσεων για να τονίσω κάποια στοιχεία που θεωρώ σημαντικά και νομίζω ότι και οι δικές σας παρεμβάσεις θα αναφερθούν σε αυτά. Η δημόσια συζήτηση μέχρι τώρα, από τότε που άρχισε η παρουσίαση της μεταρρύθμισης, επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο πρασίνισμα της ΚΑΠ. Δεν θα επανέλθω λοιπόν σε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες να το συζητήσουμε. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι λαμβάνουμε υπόψη και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό δημοσίω, λαμβάνουμε υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Γεωργία για να είναι περισσότερο πράσινη και περισσότερο ευθυγραμμισμένη με την καλή διαχείριση των φυσικών πόρων. Θέλω εδώ να τονίσω ότι από τη δεκαετία του 70-80 η χρήση των λιπασμάτων στη γεωργία μειώθηκε κατά 25% και κατά 50% η χρήση φωσφορούχων και καλλιούχων ε, λιπασμάτων. Υπάρχει λοιπόν ε, μία αλλαγή στο πνεύμα της γεωργίας και των γεωργικών πρακτικών καθώς ε, και στον τρόπο με τον οποίο η γεωργία εμφανίζεται προς τα έξω. Η σχέση μεταξύ αυτών που κάνουν οι γεωργοί και αυτών που αντιλαμβάνεται το κοινό πιστεύω ότι είναι βασική. Η ανταγωνιστικότητα, όπως έλεγε και ο Πάολο, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας περιλαμβάνει στοιχεία και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Εδώ υπάρχει μια σημαντική πρόταση που δεν την έχουμε συζητήσει πολύ από τότε που υπευλήθησαν στις 12 Οκτωβρίου ε, οι προτάσεις μεταρρύθμισης. Δηλαδή η πρόταση αυτή αφορά την οργάνωση των γεωργών και τις αγορές. Για να παραμείνει η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και για να μπορούν να παράγουν οι γεωργοί, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τις άμεσες ενισχύσεις στο εισόδημα, οι οποίες θα παγιωθούν μέχρι και το 2020 τουλάχιστον. Βεβαίως θα υπάρχει δέσμευση και για καλύτερη κατανομή αυτών των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ κρατών μελών καθώς και μέσα στο ίδιο το κράτος μέλος. Και υπάρχει και η πρόταση για το ανώτατο όριο και επίσης για τον ορισμό του ενεργού αγρότη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι περισσότερο στοχευμένα αυτά τα μέτρα. Η μεταρρύθμιση κάνει κυρίως ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα μορφή διαχείρισης των αγορών και εδώ παρεμβαίνουν όχι μόνο οι δημόσιες αρχές αλλά εμπλέκονται όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με την αγορά γεωργικών προϊόντων. Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το σύστημα παρέμβασης, δημόσιας παρέμβασης εκεί όπου είναι απαραίτητο και να διευρύνουμε την ιδιωτική αποθεματοποίηση σε όλους σχεδόν τους τομείς, ούτω ώστε να υπάρχει ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας που θα κινητοποιείται ταχαίως όταν απαιτείται. Αυτή η παρέμβαση στην αγορά δεν θα συνδέεται μόνο με τη διακύμανση τιμών στην αγορά, θα συνδέεται με οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα προκύπτει που μπορεί να έχει επιπτώσει στον α ή β κλάδο. Και γι' αυτό η πρόταση αυτή δημιουργεί πλέον ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας και μπορούμε να το κινητοποιήσουμε ταχαίως. Θα έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να το κάνει αυτό νομίζω ότι θα ελπίζω να συμφωνήσουν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σημαντικός ρόλος για την ανταγωνιστικότητα στο μέλλον θα είναι ο ρόλος της έρευνας και καινοτομίας. Θα έχουμε όμως το χρόνο να το συζητήσουμε, δεν θέλω να επεκταθώ τώρα. Να προσθέσω κάτι για το δίκτυο ασφαλείας που ανέφερα, το οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε και το οποίο θα λαμβάνει υπόψη διάφορες οικονομικές συνθήκες στους διάφορους γεωργικούς τομείς, προσαρτήσαμε ένα αποθεματικό κρίσεως, το οποίο είναι χωριστό. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη αυτή την προγραμματική περίοδο που μπορεί να κινητοποιηθεί με μια διευρυμένη ρήτρα κατεπήγοντος χαρακτήρος. Παράλληλα με αυτό, στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ προτείνουμε μηχανισμούς διασφάλισης που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη και στους γεωργούς να κινητοποιούν τον κατάλληλο προϋπολογισμό για να ενθαρρύνονται οι γεωργοί να δημιουργούν ε, ταμεία αμοιβαίας βοήθειας ή ε, δομές που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν μετεωρολογικές, κλιματικές συνθήκες που έχουν επιπτώσει στη γεωργική παραγωγή καθώς και την μεταβλητότητα των τιμών και των εισοδημάτων στις αγορές. Εκτός λοιπόν από την παρέμβαση στην αγορά θα έχουν οι αγρότες τη δυνατότητα ταμείων αμοιβαίας, ταμείων αλληλοβοήθειας που θα τους επιτρέπουν ε, να αντιμετωπίζουν την ε, μεταβλητότητα των αγορών. Θέλω να τονίσω άλλο ένα σημείο που προστίθεται σε αυτά τα δύο προηγούμενα εργαλεία. Και αυτό είναι οι οργανώσει παραγωγών. Νομίζω ότι στο μέλλον, εάν θέλουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείριση των αγορών, θα πρέπει στο κέντρο αυτή τη διαχείριση των αγορών να μην βάζουμε μια δημόσια γραφειοκρατική και δυσκίνητη αρχή, αλλά περισσότερο να βάζουμε τι οργανώσει παραγωγών. Και προτείνουμε να διευρύνουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων σε όλους τους τομείς. Να διευρύνουμε τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ισχύουν για τον τομέα των οποροκυπευτικών αυτή τη στιγμή σε όλους τους τομείς, ούτω ώστε οι γεωργοί που αποφασίζουν να οργανωθούν και να μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες δράσεις συλλογικού χαρακτήρα στην αγορά να μπορούν να την χάνουν αναγνώρισης επισήμως σε κάθε κράτος μέλος ως οργανώσεις παραγωγών ή ως ε, διεπαγγελματικές οργανώσεις. Υποχρεωτική δηλαδή αναγνώριση από τα κράτη-μέλη για όλα τα μέλη των οργανώσεων ε, των γεωργών, των οργανώσεων των παραγωγών. Προσθέτουμε και κάποιες εξαιρέσεις ε, που είναι εξυγχρονισμένες διατάξεις αντιτράστ ε, για όλους τους τομείς, όχι μόνο για τα προεκπαιδευτικά, αλλά και για τον καπνό και για τον ε, για τον ίνο, ούτω ώστε να έχουν οι οργανώσει παραγωγών ένα πραγματικό εργαλείο συλλογική δράση για να μπορούν να προγραμματίζουν την παραγωγή και να προωθούν τα προϊόντα τους και να λαμβάνουν και δράσεις συλλογικών επενδύσεων. Η δημιουργία αυτών των οργανώσεων παραγωγών θα υποστηρίζεται οικονομικά και στην αρχική φάση, αλλά και αργότερα, για να υπάρχουν προγράμματα δράσης και προγράμματα επένδυσης ή και προγράμματα διαχείρισης της αγοράς. Και στο μέλλον, όσο θα προχωρούν τα εργαλεία διαχείρισης των αγορών, Σιγά σιγά θα μπορεί να στρέφεται αυτό γύρω από τις οργανώσεις παραγωγών, εφόσον βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το μέτρο αυτό. Οι οργανώσεις παραγωγών θα μπορούν να κάνουν τα πάντα, θα έλεγα. Προγραμματισμό της παραγωγής, επενδύσεις. Το μόνο που δεν θα μπορούν θα είναι το να καθορίζουν τις τιμές ή να καθορίζουν ποσοστώσεις. Εκτός αυτού, Μπορούν όλα τα άλλα να τα κάνουν με συλλογικό τρόπο και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο ο ρόλος των οργανώσεων ενισχύεται κατά πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να τονίσω σήμερα, γιατί αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει πολύ. Παράλληλα με τις άμεσες πληρωμές, με τις άμεσες ενισχύσεις, αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν στους αγρότες να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και η ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή κατά τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να κερδίσει τη θέση που της αξίζει στην παγκόσμια αγορά. Και η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εξεταστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν τα μέσα για την αηφοροδιαχείριση και υπάρχουν και όλα αυτά τα εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη την καινοτομία και την έρευνα στη γεωργία και θα δίνουν τη δυνατότητα στους γεωργούς να παράγουν καλύτερα με τρόπο περισσότερο προσαρμοσμένο σε αυτά τα οποία θέλει η κοινωνία και η αγορά. Αυτά ήθελα να σας τονίσω και ελπίζω ότι στις παρεμβάσεις σας θα αναφερθείτε σε αυτά τα στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε μέσα στα προσεχή χρόνια, στην προσεχή περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γκαριτζάνο τώρα. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, λέει ο κύριος Ζων Λάιτνερ, Πρόεδρος της ΚΟΠΑ, κύριε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την, την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου για την οργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής συζήτησης. και λαμβάνω το λόγο εκ μέρους ε, όλων των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτά τα οποία θα γίνουν στο μέλλον στη Γεωργία, θα πρέπει ε, να φροντίσουμε ε, την παγκόσμια αυξανόμενη ζήτηση για είδη διατροφής και τη σπάνιδα των πόρων καθώς και την αλλαγή του κλίματος. Είναι πολλές οι προκλήσεις για τη γεωργία. Είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη γεωργίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάπτυξη στο πλαίσιο της τωρινής κρίσης στην Ευρώπη είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Ο τομέας της γεωργίας και ο τομέας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός και την περασμένη εβδομάδα στο G20 συζητήθηκε το θέμα της αυξανόμενης παραγωγικότητας της γεωργίας και της ε, ασφάλειας, ε, της επιστηστικής ασφάλειας που πρέπει να προωθήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής μας ανησυχεί. τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται δεν είναι μέτρα που θα βελτιώσουν τη γεωργία και την προστασία του κλίματος. Η γεωργοί είναι η καλύτερα, αυτοί που είναι καλύτερα σε θέση να βελτιώσουν την παραγωγή και να προστατεύσουν το κλίμα. Δεν θα πρέπει όμως ε, να εμποδίζεται η παραγωγικότητα των γεωργών γιατί αυτό θα είναι εις βάρος της επιστημιστικής ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της το θέμα που αφορά την οικολογική ανάπτυξη, αλλά δεν έχει λάβει υπόψη το ε, τμήμα το οποίο αφορά την παραγωγικότητα της γεωργίας. Η πρόταση του ε, να αποσύρεται από την παραγωγή το 7% των γεωργικών γεών είναι μια πρόταση η οποία μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους. Δεν έχει νόημα μια τέτοια πρόταση. Προσπαθούν οι κυβερνήσεις ε, να χρησιμοποιήσουν βιοενέργεια και βιοαποδομήσιμα υλικά και εμείς αυτά θέλουμε να τα συνδυάσουμε με βιώσιμη γεωργία. Θα πρέπει ε, ε, να λυθούν υπόψη οι ανάγκες των γεωργών, των οποίων οι δαπάνες αυξάνονται ενώ παράλληλα θέλουν να εξασφαλίσουν μέσα διατροφής για τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να μην εξαρτάται η Ευρώπη από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν οι αγρότες και πρέπει οι αγρότες να συνεισφέρουν ε, στην προστασία του κλίματος και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας ε, την γεωργική παραγωγή. Η δική μας απάντηση είναι ότι θέλουμε να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη. Η Επιτροπή μιλά για την νομιμοποίηση της ΚΑΠ και για τα μέτρα που προτείνονται για τις άμεσες πληρωμές εμείς όμως πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να ζούμε σε ένα ε, κόσμο με ασφάλεια και αν θέλουμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη σε μεγαλύτερη απασχόληση και μεγαλύτερη ανάπτυξη, η κοινή γνώμη σαφώς θα αναγνωρίσει ότι το κόστος της ΚΑΠ είναι λιγότερο από 1% ε, ε, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει η ανάπτυξη της υπαίθρου να αποτελεί τμήμα της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020 και παράλληλα να οδηγεί σε έξυπνη ανάπτυξη. Ένα περαιτέρω πρόβλημα το οποίο έχουμε με την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι δεν υπάρχει καμία απλοποίηση. Υπάρχουν οι προτάσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση, για το πρασίνισμα της γεωργίας, διατάξεις που κάνουν το σύστημα πολύ λίγο διαφανές για την κοινή γνώμη και δεν δίνουν την δυνατότητα φιλικής αντιμετώπισης από τους αγρότες. Υποστηρίζουμε το ε, σύστημα των άμεσων πληρωμών σε ενεργούς αγρότες, αλλά καλύτερα θα ήταν να υπήρχε κάποιο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη, που θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ποιον θεωρούν ενεργό αγρότη και ποιον όχι. δεν πρέπει η ΚΑΠ να φύγει αυτούς οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να εξυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους. Η Επιτροπή μιλά για νέα κατανομή των ε, άμεσων ε, πληρωμών ε, και ε, αυτό μας βρίσκει σύμφωνους εφόσον υπάρχει δίκαιη μεταχείριση για όλους τους αγρότες και εφόσον λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα οποία από την αρχή τονίσαμε ως περισσότερο σημαντικά. Το να υπάρχει ένα καταποκοπή ποσό σε όλα τα κράτη-μέλη δεν θα είναι για όλους τους αγρότες ε, σωστό, γιατί θα χρειάζονται περισσότερη ευελιξία και περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα νέο σύστημα καταποκοπής πληρωμών και θα πρέπει οι αλλαγές να εισαχθούν ε, σταδιακά και όχι με βάση το 40% τον πρώτο χρόνο που προτείνει η Επιτροπή, γιατί αυτό θέτει μεγάλη επιβάρυνση ήδη από την αρχή και δεν αφήνει χρόνο προσαρμογής στους αγρότες. Θέλουμε να υπάρχει σωστός βαθμός σύνδεσης των πληρωμών και δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το διαχωρισμό που προτείνει η Επιτροπή για τις διάφορες περιφέρειες ε, για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Αυτό αποτελεί... Αυτό προσθέτει ένα χαρακτήρα πολυπλοκότητα στο σύστημα και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τις ε, ιδιαίτερα βεβαρημένες περιοχές. Θα θέλαμε να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις για την πράσινη ανάπτυξη και εμάς μας ανησυχεί το πώς θα λειτουργήσουν, θα λειτουργήσουν στην πράξη αυτές οι προτάσεις στρατηγικής. Υπάρχουν βέβαια στο δεύτερο πυλώνα και κάποια σημεία τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους. Οι θεματικές, παραδείγματος χάρη προσεγγίσεις, μας βρίσκουν ε, ε, σύμφωνους. Και το θέμα της καινοτομίας επίσης μας βρίσκει σύμφωνους και ελπίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι σχέσεις καινοτομίας θα οδηγήσουν σε ένα μέλλον όπου η έρευνα θα βοηθήσει την γεωργία και αντιστρόφως. Η σταθερότητα είναι ένα σημαντικό σημείο της διατροφικής ασφάλειας και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε μηχανισμούς του παρελθόντος. Θέλουμε όμως οι μηχανισμοί να δίνουν γρήγορες απαντήσεις σε περίπτωση κρίσεως και να επιφέρουν σταθεροποίηση. Τα αποθεματικά κρίσεις της Επιτροπής θα πρέπει εδώ να μπορούν να διατεθούν καταλήλως. η γεωργία θα πρέπει να βοηθά τον ασφαλή εφοδιασμό και είμαστε πεπισμένοι ότι η απάντηση της Επιτροπής στις προκλήσεις που τίθενται μπορεί να βελτιωθεί. Θα χρειαστούν συζητήσεις αλλά πιστεύουμε ότι το μέλλον της ΚΑΠ μπορούμε να το αποφασίσουμε γνωρίζοντας βέβαια και τον προϋπολογισμό ο οποίος θα διατεθεί. Θέλουμε από κοινού να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα συνεισφέρει ε, στο να γίνει ο τομέας της γεωργίας ένας τομέας αποδοτικός που θα είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τη σημασία της κοινή γεωργικής ε, πολιτικής στο μέλλον. Μακάρι να λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο καλά και σε άλλους τομείς όπως λειτουργεί στον τομέα της γεωργίας. Δεν θα είχαμε τότε τη σημερινή οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γκέρτ και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον ε, Πάολο Μπρούνι που είναι πρόεδρος της ε, Κοτζέκα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Σαβίτσκι. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον Πάολο Ντεκάστρο και τον Επίτροπο Τσόλος, καθώς και όλους τους ευρωβουλευτές με τους ε, προσκαλεσμένους αυτής της ημέρας. Εγώ θα ήθελα από πλευράς ε, Κοτζέκα, δηλαδή από πλευράς ε, συνεταιρισμών ειδών διατροφής όπου συμμετέχουν 38.000 ε, εκμεταλλεύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τη συνεισφορά μου από πλευράς Κοτζέκα. Στις 12 Οκτωβρίου η Επιτροπή προέβησε μία ανακοίνωση. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Επίτροπος Τσόλος, θα ήθελα να σταθώ σε θέματα αγοράς καθαρά και ανταγωνιστικότητας. Εμείς, ως προς αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ χρόνο, γιατί θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι επιχειρήσεις μας, οι συνεταιρισμοί μας, έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι προδιαγραφές ασφάλειας και ο σεβασμός του περιβάλλοντος δεν είναι τα ίδια. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο για εξοκοινωτικές εκμεταλλεύσεις να παράγουν με χαμηλότερο κόστος. Θα πρέπει λοιπόν με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να ορίσουμε μηχανισμούς που επιτρέπουν στις δικές μας εκμεταλλεύσεις να είναι ανταγωνιστικές για το μέλλον της γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της απασχόλησης που δυστυχώς ε, λίγες φορές θυμόμαστε, γιατί μιλάμε για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας περισσότερο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατροφική αλυσίδα και ο γεωργικός τομέας απασχολούν έναν ανά έξι εργαζόμενους σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας. Μιλάμε δηλαδή για υψηλό απασχόληση στην Ευρώπη. Ένα στους έξι εργαζόμενους. Πολλοί μίλησαν για την ανάγκη μεγαλύτερης παραγωγής, μίλησαν για την ανάγκη ανάπτυξης που απορρέει και από τις προβλέψεις της ΦΑΟ για τα επόμενα έξι χρόνια. Σε αυτό το θέμα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα αντικειμενικά στοιχεία τα οποία για τις πορές μας δείχνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι κάτω από 1%. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει έρευνα και να προβληθεί καινοτομία έτσι ώστε να παράγουμε περισσότερο. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια άλλη πτυχή που κατά την άποψή μου εντάσσεται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, γιατί το να είναι ανταγωνιστική μια επιχείρηση σημαίνει ότι έχει καλή απόδοση στη διατροφική αλυσίδα. Ο πρώτος κρίκος της διατροφικής, διατροφικής αλυσίδας είναι η γεωργία. Εάν δούμε όμως τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε ότι στη γεωργία πάει το μικρότερο μέρος του κέρδους, δηλαδή λίγα λεπτά του ευρώ που μπαίνουν στη τσέπη του γεωργού. Άρα θα πρέπει να προβούμε σε μία εξισορρόπηση. Υπάρχει και το φόρμ της ανταγωνιστικότητας που απασχολεί τον Αντώνιο Ταγιάννη, τον Επίτροπο, που ασχολείται με αυτό το θέμα, αλλά όπως έλεγα, λίγες μέρες πριν ε, στον κύριο Τσόλος, ο οποίος μετέβη στη Ρώμη, πιστεύω ότι και, το, και η πολιτική της ΚΑΠ θα πρέπει να επανισορροπήσει την διατροφική αλυσίδα και το, το γεγονός ότι το Φόρουμ Ανταγωνιστικότητας προσπαθεί να παράγει αποτελέσματα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ. Λαμβάνω υπόψη όσα προβλέφθηκαν από την πρόταση μεταρρύθμισης έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε διεπαγγελματικά. Και αυτό μας οδηγεί στο σωστό δρόμο, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τον τρόπο και την τυπολογία αυτών των οργανώσεων. E και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα βήματα και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς εξελίσσεται και ο τομέας των οποροκυπευτικών. Στον τομέα των οποροκυπευτικών οι επαγγελματικές οργανώσεις διαθέτουν πλήρη ελευθερία για την εμπορία των προϊόντων. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα που αφορά τις οργανώσεις των παραγωγών. Εμείς στην Κοτζέκα πιστεύουμε ότι ένα ιδεώδες μοντέλο και πρότυπο θα αφορούσε μία συνεταιριστική μορφή. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια πραγματική, ένα πραγματικό εγχείρημα ουσίας θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στα ε, μέσα διαχείρισης της κρίσης που υπενθυμίστηκαν εδώ και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσουν ε, απαράβατο στοιχείο της σκέψης μας. Ο κύριος Ντες, όταν άρχισε να μιλά για αυτά τα μέσα διαχείρισης της κρίσης, μιλήσαμε για τη γεωργία του μέλλοντος, που δεν θα είναι ίδια με εκείνη του παρελθόντος. οι κρίσεις θα είναι ολοένα και διονγκούμενες και επαναλαμβανόμενες εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο Γεωργός δεν θα πρέπει να χάνει το εισόδημά του. Θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις κρίσεις έτσι ώστε για το μέλλον να αποτελούν ένα στοιχείο που να μπορούν να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό αφορά και τον Επίτροπο Τσόλος και την δική σας Επιτροπή και το Συμβούλιο. Υπάρχει ένα χρονικό καθαρά στοιχείο για τη διαχείριση της ε, κρίσης. Το 2012 υπάρχει ένα ανοιχτό πρόβλημα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση των παραγωγικών τάξεων και ιδιαίτερα εκείνων που παράγουν οποροκυπευτικά που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά δεν έχουμε την οριστική απόφαση αυτών των ε, ε, πόρων. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω κατανοήσει την ε, πλαισίωση αυτή. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι να εκφράσω μία ευχή. Ήδη έγιναν δύο συναντήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Επίτροπος μας είπε ότι στις 19 Δεκεμβρίου η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τον κύκλο αντιπαραθέσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι οι θέσεις είναι σαφής και ήρθε η ώρα, όπως είπα και χτες τον κύριο Κάπουλα Σάντος, ότι θα πρέπει να ε, συγκλίνουμε ως προς τις ε, θέσεις επιτάπητος. Αυτές οι αντιπαραθέσεις έχουν ένα νόημα, να κατανοήσουμε τις διαφορετικές θέσεις και να φτάσουμε σε μία κοινή θέση με βάση τις συγκλήσεις που προβλέπονται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάολο, αναφέρθηκε στο μέλλον εμπολίσει και νομίζω ότι οι νέοι γεωργοί ανησυχούν ιδιαίτερα. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Γιώρη Μπέκε που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Νέων Γεωργών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Υπουργέ Σαβίσχη. Κύριε Δεκάστρο, κύριε, Υπουργέ, κύριε, Commission, ε, ε, κύριε Πίτροπε, συγγνώμη και όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία που οργάνωσε τη σημερινή συνάντηση και θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του 1,8 εκατομμυρίων νέων αγροτών, τους οποίους εκπροσωπεί η ΣΕΖΑ. Οι φιλοδοξίες και οι προκλήσεις του μέλλοντος απαιτούν μια νέα ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική. Και για να ανταποκριθούμε σε αυτές ε, τις νέες προκλήσεις, ε, η κοινή αγροτική πολιτική χρειάζεται ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό. Η γεωργική παραγωγή βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όχι μόνο σε υλικά, αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Και όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, εδώ υπάρχει μία απειλή για τη γεωργία, γιατί υπάρχει ο πληθυσμός που απομακρύνεται από την Ήπεθρο και δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι που θέλουν να μπουν στον τομέα της γεωργίας. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια ηλικιακή κρίση η γεωργία στην Ευρώπη και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όταν μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για επενδύσεις στο μέλλον και η ΚΑΠ πρέπει να επενδύσει στην γεωργία του μέλλοντος και στα αγροκτήματα του μέλλοντος και πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα. Η ΣΕΖΕ συμφωνεί για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα που πρότεινε ο Επίτροπος μέτρα υπέρ των νέων αγροτών. Συμφωνούμε με τις άμεσες ενισχύσεις του τους νέους γεωργούς τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την ε, εγκατάστασή τους, γιατί αυτό αναγνωρίζει τον ευπαθή χαρακτήρα των νέων αγροτών, γιατί υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Θα θέλαμε όμως ε, να ενισχυθεί κάπως η πρόταση σε κάποια σημεία της, γιατί πρέπει το μέτρο αυτό να είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει ένα ελάχιστο 2% του κάθε εθνικού κονδυλίου να χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί αυτό το μέτρο. Και για την εφαρμογή αυτού του μέτρου χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο κρατών μελών για να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των νέων αγροτών όσον αφορά το 2011 ως έτος αναφοράς για να υπολογιστεί ε, ε, ως έτος αναφοράς για τα έτη από το 2014 και μετά αυτή είναι μια διάταξη που δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για τους μελλοντικού νέους αγρότες που θα θέλουν να μπουν σε αυτό το τομέα και θα πρέπει από το 2014 και μετά να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τα δικαιώματα των νέων αγροτών ε, που θα είναι νέο εισερχόμενοι στη Γεωργία. Για το δεύτερο πυλώνα χαιρετίζουμε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής όσον αφορά τους νέους αγρότες, ιδιαίτερα τη συγχρηματοδότηση που θα παρέχεται κατά προτιμησιακό τρόπο στους νέους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανανέωση των γενεών στη γεωργία, βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη και για βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Η ΣΕΖΑ υποστηρίζει ένα πιο πράσινο πρώτο πυλώνα, Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι ο γεωργικός τομέας είναι ο πιο πράσινος τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για να φτάσουμε ε, τις δεσμεύσεις των αγροτών και για να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εθελοντικό το πρασίνισμα και τα μέτρα τα οποία προτείνονται δεν δίνουν απάντηση στις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις ούτε στην πολυμορφία των Ευρωπαίων γεωργών. Γι' αυτό προτείνουμε μέτρα τα οποία θα πληρούν τις ανάγκες βιοπικιλότητας και κλίματος καθώς επίσης και τις ανάγκες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα πολλά ε, μέτρα τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση των υδατικών πόρων και τη διαχείριση του εδάφους ε, και μέτρα αύξησης της αποτελεσματικότητας της γεωργίας συστήματα που θα βασίζονται σε καλλιέργειες οσπρίων, ε, σε ζώνες διαχωρισμού καλλιεργιών, και με αυτά τα μέτρα θα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και θα επωφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να τονίσω ότι οποιοδήποτε σταθερό ποσοστό οικολογικών περιοχών σε επίπεδο αγροκτημάτων θα είναι αντιπαραγωγικό και δεν απαντά στις πραγματικές προκλήσεις για την αηφόρο διαχείριση. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αγρανάπαυση και μόνο, πράγμα το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με, την, με το αίτημα για μεγαλύτερη παραγωγή ειδών διατροφής. Συνεχίζουμε τις εσωτερικές μας συζητήσεις για να διαμορφώσουμε την τελική μας θέση. Πάντως η ανάγκη για κερδοφόρο τομέα, κερδοφόρο γεωργικό τομέα θα πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Τονίζω ότι θέλουμε σημαντικά εργαλεία για την ανανέωση των γενεών στη Γεωργία, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο να σας μιλήσω σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Τέσσερα λεπτά ο κάθε μιλητής. Αν το σεβαστούν όλοι αυτό θα μπορέσουν να μιλήσουν περισσότεροι. Καπούλας και Σάντος ο πρώτος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην εκτίμηση της πολιτικής μου ομάδας προς την Πολωνική Προεδρία, διότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μία από τις πολλές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, ο οποίος βρίσκεται πολύ συχνά στο Κοινοβούλιο και είμαι σίγουρος ότι με την ανταλλαγή αυτή απόψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Ως Ευρωβουλευτής και συντονιστής της Σοσιαλιστικής Ομάδας έχω σαφείς απόψεις για αρκετές πτυχές της μεταρρύθμισης που παρουσίασα δύο χρόνια πριν σε ένα δημόσιο έγγραφο, έγγραφο και χαίρομαι διότι η Επιτροπή ε, ενσωμάτωσε πολλές προτάσεις στο εγγραφό της. Άλλες βεβαίως δεν εισήχθησαν, αλλά θα προσπαθήσουμε να τις εισαγάγουμε μέσα σε αυτή τη ε, διαπραγμάτευση. Δεν θα ήθελα να εκφράσω απόψεις ο συντονιστής, θα ήθελα να ακούσω τις υποδείξεις και τις επικρίσεις οι οποίες θα με βοηθήσουν στη σύνταξη της έκθεσής μου. Καταρχήν, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι μετά τις 12 Οκτωβρίου η Επιτροπή επικρίθηκε εσφαλμένα πολλές φορές, γιατί τονίζουμε τις αρνητικές πλευρές πρότασης και ξεχνάμε τις θετικές. Η Επιτροπή ενέχει και θετικά στοιχεία και άλλα που θέλουμε να βελτιώσουμε. Θα θέλαμε όμως να σταθούμε σε στοιχεία που δεν μας ικανοποιούν τόσο πολύ. στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου και στον κανονισμό άμεσων πληρωμών δεν θεωρούσα ότι θα είχε την κατανομή των εθνικών κονδυλίων στο παράρτημα 2 και στο παράρτημα 3, γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδίνωση του θέματος. Θα ήθελα να έχει επιλέξει τα κριτήρια και από την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων να οριστούν τα εθνικά κονδύλια, η εθνική συμμετοχή όπως γινόταν μέχρι τούδε. Επίσης, έχουμε και μία παράλληλη συζήτηση σε σχέση με το γενικό προϋπολογισμό ως προς την ΚΑΠ. Και ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το greening το πρασίνισμα. Όλοι θεωρούμε ότι αυτό το σκέλος της ΚΑΠ είναι πολύ σημαντικό για την ε, αποδοχή της από την κοινωνία. Θα πρέπει όμως αυτό να αποσαφινιστεί καλύτερα από την Επιτροπή διότι αποτελεί έναν πυλώνα πολύ σημαντικό για την ΚΑΠ θα πρέπει να εξεύρουμε μία λύση που να είναι πιο ικανοποιητική για όλους, όπου να σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά να λάβουμε υπόψη και το σκέλος της ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισελ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος ολόκληρου του Κοινοβουλίου επεφορτίστην να συγγράψω μια αναφορά, μια έκθεση για την κοινή οργάνωση των αγορών γενικότερα και θέλω να χαιρετήσω την εργασία της Επιτροπής και του Επιτρόπου που μας έδωσαν τις δυνατότητες ε, οργάνωσης ε, των οργανώσεων των γεωργών μπροστά στην ε, στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Τώρα, το θέμα είναι γιατί όλα αυτά. Δεν αρκεί να υπάρχει καλή οργάνωση των παραγωγών με επαγγελματικές οργανώσεις κλπ. Πρέπει παράλληλα αυτό να εξυπηρετεί κάτι πραγματικά στην αγορά. αν και δεν πρόκειται να καθορίζει τη μέση η οργάνωση των Γεωργών, αν και στην περίπτωση της ΚΟΠΑ και ΚΟΖΕΚΑ, στο παρελθόν το έπρατε. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα οργανωθούν όλα αυτά. Τώρα για την ανταγωνιστικότητα και το δίκαιο αυτής. Πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την εφαρμογή του άρθρου 101 της συνθήκης και του 40 Παλιά υπήρχαν κοινέ οργανώσεις αγορών που σήμερα πρέπει να επαναδιοργανωθούν. Η κοινή οργάνωση της αγοράς που παρουσιάζεται σήμερα πρέπει να ανταποκριθεί, να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση που την αναφέρουμε και σε μια έκθεση του Κοινοβουλίου πριν από μερικούς μήνες, το 1995, ο κύκλος εργασιών του γεωργικού τομέα ήταν 475 δισεκατομμύρια εξών 31% επέστρεφαν, ήταν έσοδα των γεωργών. Ενώ το 2008 171 και πολύ μικρότερο ποσοστό στους γεωργούς. Αυτές οι διαφορές δείχνουν ότι έχουν υποβεληθεί όλοι εκτός από τους παραγωγούς. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα θα μπορούμε με τον πρώτο και τον δεύτερο πυλό να βάζουμε όσα χρήματα θέλουμε, αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό. Θα τους ακούσω όλους για να βρούμε μια λύση σε συνεργασία φυσικά και με τον Επίτροπο και τις υπηρεσίες του. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συμπρόεδρε, συνάδελφοι, εμπειρογνώμονες. Και εγώ ευχαριστώ τον Επίτροπο Τσόλος για όσα μας παρουσίασε. Τεράστιος φόρτος εργασίας, 600 σελίδων. Πώς θα εφαρμοστούν όμως όλα αυτά τα μεμονωμένα κτήματα. Θα ήθελα να τονίσω μερικά, μερικές λεπτομέρειες όπου νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό το 7% ο κανόνας που αναφέρθηκε. Είπατε ότι δεν αποκλείει ορισμένα στοιχεία από ό,τι ίσχυε στο παρελθόν. Αλλά εάν δω στη χώρα μου το 70, τη δεκαετία του 70. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ήδη 10% χορηγείται, πιο 7%. Και τώρα ζητάμε από το μεμονωμένο αγρότη να εφαρμόσει έναν κανόνα που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Κάποιος που έχει μεγάλα κτήματα δεν έχει το ίδιο πρόβλημα με κάποιον που έχει μικρότερα. Άμα δούμε τους αριθμούς καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι πληρώνουν υψηλά ποσά για κτήματα που δεν διαθέτουν ή που δεν καλλιεργούν μάλλον καλλιεργούν 10 εκτάρια για να πληρώσουν τα υπόλοιπα 3,5 που έχουν παγώσει, που απαγορεύεται η καλλιέργειά τους. Αυτά δεν είναι λύσεις, είναι μπαλώματα. Όταν σε κάποια περιφέρεια έχουμε γεωργούς με κτήματα που δεν καλλιεργούνται μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό αφορά μόνο μικροκαλλιεργητές. Παραδείγματο χάρη. Είναι γνωστό ότι και κοντά στα ορυχεία υπάρχουν καλλιεργήσιμες γέες. Οι αγρότες λοιπόν τι κάνουν. Βάζουν οποροφόρα δέντρα όποτε είναι ανώμαλο το έδαφος και αυτό το όριο των τριών εκταρίων είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, να γίνει 15 ή 20 εκτάρια, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και πρέπει να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι συμβιβασμοί και άλλοι υπολογισμοί για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικές ζώνες πτωχότερες από άλλες, υποδέστερες, όπου πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις για τους γεωργούς τους. Επίσης ξέρουμε ότι μερικά κράτη όπως η Βαλγαρία καλύπτονται από τον δεύτερο πυλώνα. Ενώ τώρα θα πρέπει ένα τμήμα των γεών τους να περάσει στον πρώτο λένε μέχρι και 20%. Προηγουμένως επρόκειτο για συγχρηματοδότηση. Τώρα τι θα κάνουν με τον πρώτο πυλώνα. Νομίζω κύριε Επίτροπε ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε γιατί και εσείς είστε διατεθειμένος. Και αυτό θα είναι το κύριο καθήκον των συζητήσεων και εδώ στο Κοινοβούλιο και στη συνεργασία με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στις προσπάθειές μας ε, και τους αγρότες, ούτως ώστε να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. Ευχαριστούμε κύριε και κύριε Υπουργέ, για αυτή τη ε, διοργάνωση της σημερινή συνεδρίασης, γιατί νομίζω ότι είναι θετικό τα θεσμικά όργανα από εκείνο να προσπαθούν να βρίσκουν λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Ρικιέτσιο εκπρόσωπο των Συμβουλίων Γεωργών στη Δανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ τη δυνατότητα που μου δίνετε να λάβω το λόγο σήμερα. Και θα ήθελα ε, ε, να μιλήσω εκ μέρους των παραγωγών στη Δανία που εκπροσωπούν και μεγάλο μέρος ε, του εξαγωγικού εμπορίου. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα γεωργικά προϊόντα σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες και παρατηρούμε ότι οι αγρότες θα πρέπει να συνεχίσουν να παράγουν και να αυξάνουν την παραγωγή τους χωρίς να αυξάνεται παράλληλα και η δυσμενής επίπτωση στο περιβάλλον, πράγμα το οποίο αποτελεί μια επιπλέον δυσκολία. Θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη χωρίς να τα μετατοπίζουμε σε χώρες του τρίτου κόσμου. Άλλη μια πρόκληση λοιπόν για τη Γεωργία. και παράλληλα θέλουμε με τη Γεωργία να προωθήσουμε και μια πολιτική ανάπτυξη για τις χώρες της Ευρώπης στο μέλλον. Για τις ενισχύσεις υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης και ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με την χρηματοδότηση που έχουμε στη διάθεσή μας και με τα κριτήρια ε, και τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε έναντι του περιβάλλοντος. θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να εφαρμόσουν στην πράξη σε κάθε κράτος μέλος τα μέτρα τα οποία προτείνονται για το γάλα και τα οποροκυπευτικά παραδείγματο χάρη, χωρίς ε, να αυξάνουμε τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χουάν Κορπόραν έχει το λόγο από έναν Ισπανικό συνεταιρισμό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οργάνωση που εκπροσωπώ ε, περιέχει 4.000 συνεταιρισμούς ε, για, στον τομέα του ίνου, του γάλακτος, των οποροκυπευτικών. Μιλάμε για έσοδα 20 δις και απασχολούν ένα εκατομμύριο αγορότες ε, και αποτελούν το 50% της τελικής παραγωγής. Ε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τα θετικά στοιχεία, τα οποία είναι πολλά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της διατροφικής αλυσίδας. Θεωρούμε ότι ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η πυγμή των γεωργών στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας, αλλά θεωρούμε ότι τα μέτρα δεν είναι αντίστοιχα. Η Κομισιόν λέει ότι ε, αναγνωρίζονται όλοι οι τιμείς. Ο κανονισμός το επιτρέπει γιατί ο κανονισμός 79 2000 το επιτρέπει. Υπάρχει όμως ένα θέμα που είναι η παρέκταση του κανονισμού και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Δεν υπάρχει όμως ένα κατόφλι στην πρόταση δεν γίνεται λόγος για τα τεχνικά και ανθρώπινα μέσα για να επιτύχουμε τους στόχους. Με την παρούσα πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσαν δύο αγρότες να έχουν ένα γραφείο και έναν χι αριθμό παραγωγών. Στο άρθρο 106 της πρότασης θα πρέπει να ορίσουμε κοινούς κανόνες εμπορίας με βάση το, ανθρώπινο δυναμικό. Οι οργανώσεις παραγωγών που έχουν ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να ορίσουν τιμές, να ορίσουν καλύτερα τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης. Αν λοιπόν δεν βελτιωθεί το άρθρο 106, δεν θα μπορέσουμε να ορίσουμε καλύτερα την προσφορά. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει μία βελτίωση και στον τομέα του γάλακτος. Θα θέλαμε λοιπόν να προχωρήσει η Κομισιόν με το άρθρο 106. Επίσης, με βάση το άρθρο 125α και β δεν ορίζονται επαρκώς τα οποροκυπευτικά. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί στη βασική νομοθεσία έχουν αρθεί αυτά τα δύο ε, άρθρα, όπως ισχύουν στον τομέα του ίνου, της ζάχαρης των οποροκυπευτικών και ούτω καθεξής. Έγινε λόγος για κατεξουσιοδότηση πράξης, αλλά βλέπουμε ότι δεν αντικατοπτρίζονται αυτό το, τα δύο άρθρα. Επίσης το κάπινγκ μας απασχολεί ιδιαίτερα γιατί μία, ένα συνεταιρισμός λαμβάνει ένα εκατομμύριο ευρώ με μία ενία καταβολή. Αλλά το κάπινγκ δεν θα πρέπει να αφορά μόνο του συνεταιρισμούς. Θα πρέπει να δίδεται και στους μικρούς γεωργούς και θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία για αυτούς τους μικρούς γεωργούς ή εκμεταλλεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάντσο Σάντσες έχει το λόγο. Bonjour. Bonjour. Ευχαριστώ. Από την οργάνωση Βία Καμπεσίνα Ο κύριος Σάντσες ε, δυστυχώς χρειάστηκε να φύγει σήμερα το πρωί για την Ισπανία, οπότε θα λάβω εγώ το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βία Καμπεσίνα έχει παρουσία σε 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα εξ να κάνω μια δήλωση. Ο κύριος Σαβίκ, ε, ε, κύριος Δεκάστρο, ε, που είναι εδώ παρόντες, πρέπει να ακούσουν ότι μας εκπλήσει ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε αυτή η συζήτηση. Παρουσιάζεται αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση με τις τομεακές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά εδώ και 45 λεπτά μόνο την κόπα Κοζέκα Σέζα ακούσαμε, η οποία κατά κανένα τρόπο δεν εκπροσωπεί όλους τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Γεωργίας ε, από το 1987 μα ακούει. Σήμερα το πρωί έγινε μια κρόση των γεωργικών οργανώσεων ε, με την ΚΟΠΑ και την Ευρωπαϊκή ε, Οργάνωση Βία Καμπεσίνα με ίσο χρόνο εργασία. Δεν υπάρχουν επαρκή δημοκρατικά δικαιώματα για μας. Το μονοπόλιο εκπροσώπηση, είτε για πολιτικούς είτε για συνδικαλιστικούς λόγου μα θυμίζει σκοτεινές εποχές του 20ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι είχε ανοίξει τη συζήτηση της ΚΑΠ στην κοινωνία των πολιτών και χαρήκαμε που άνοιξε και συμπεριέλαβε και την κοινωνία των πολιτών και όντως πρέπει να ανοίξει ο διάλογος και να μην αποτελεί μια κλειστή συζήτηση. Ζητούμε από τον Πρόεδρο της ε, Επιτροπής Γεωργίας ε, του Κοινοβουλίου και από την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου να διοργανώνουν συζητήσει πλουραλιστικέ που θα εκπροσωπούν την πολυμορφία της κοινωνία. Για σήμερα το απόγευμα, και ε, λυπάμαι γι' αυτό, η προσωπική μου και συνδικαλιστική ε, δεοντολογία μου υπαγορεύουν να φύγω από την αίθουσα γιατί είναι ιερή η νόμη της δημοκρατίας. Καλό τους συμμετέχοντες που θέλουν να παραμείνουν στην αίθουσα να λάβουν υπόψη τις θέσεις μας, την οποία θα αφήσουμε γραπτός στο τραπέζι εδώ αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Σας Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την εκδήλωση ανεξαρτησίας που κάνατε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι να οργανώνουμε ευρωπαϊκές συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ. Η δήλωσή σας θα ληφθεί δεόντως υπόψη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Σουηδία, τον κύριο Χόλστρομ δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ομοσπονδία Σουηδών Αγροτών Λερεφ εκπροσωπεί 170.000 γεωργούς που διαθέτουν κτήματα και δάση καθώς και εκπροσωπεί 28 συνεργατικές οργανώσεις. Η ΕΛΕΡΕΦ θα ήθελε να υπάρξει μια κοινή αγροτική ε, πολιτική που να προωθεί τη γεωργία με βιώσιμο και ηθικός σωστό τρόπο. Χαιρόμαστε που οι προτάσεις σας της Κομισιόν αναγνωρίζουν τη σημασία της γεωργίας για την παραγωγή τροφίμων στην Ένωση. Η πρόταση είναι μια σωστή βάση για τη συνέχιση της ΚΑΠ και υποστηρίζουμε την προσπάθεια της Κομισιόν να γίνει πιο βιώσιμη η ΚΑΠ. Αλλά αν και υποστηρίζουμε και κατανοούμε την ανάγκη μιας πρασινότερης ΚΑΠ, νομίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί πρασίνισμα που να ισχύει ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ευρώπη, οι καλλιεργήσιμες ποικιλίε μπορεί με τα μέτρα αυτά να καταλήξουν σε περισσότερη γραφειοκρατία όπως στη δική μου χώρα. Επίσης πιστεύουμε ότι, ότι ε, το πρασίνισμα της ΚΑΠ δεν αρκεί για να γίνει βιώσιμη αυτή. Αντί για αυτά τα μέτρα θα θέλαμε να υπάρξει ένα πρασίνισμα που να δημιουργεί πράσινη ανάπτυξη. Και ένας τρόπος θα ήταν οι γεωργοί να εφαρμόζουν τα πρασινομέτρα αυτομάτως και έτσι να προωθούν ενεργά την βιώσιμη γεωργία, πράσινο γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριος Ιούζη Κορσικόφσκι. Σας ευχαριστώ Υπουργέ για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. Χαίρομαι γιατί μπορεί να γίνει μια πραγματική ε, συζήτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές που υποβλήθηκαν από τον Επίτροπο δεν είναι ακριβώς αυτό που αναμενόταν. διότι δεν μιλάμε για μία μακρόπνοη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτό επιθυμούσαμε και θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε σωστούς όρους ανταγωνισμού για τον Ευρωπαίο Γεωργό με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό όμως που αντιμετωπίζουμε και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι εστιάζεται την ε, προσοχή στους μεγάλους δικαιούχους σε σχέση με τους μικρούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει άλλη μεταβατική περίοδο για τις άμεσες πληρωμές και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση Αυτό θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις ανταγωνισμού μέσα στην ενιαία αγορά. Δεν υποστηρίζουμε τον άδικο, τα άδικα αυτά μέτρα ανταγωνισμού κατά των Πολωνών αγροτών αλλά νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος των 12 νέων κρατών που βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από τα παλαιότερα 15 κράτη. Θα πρέπει να επανεξεταστούν ορισμένα μέτρα, να δούμε πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα. Και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, δεν μπορεί να γίνει επανακατανομή. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις παλαιότερες αρχές. Τώρα όμως και με τα νέα κράτη-μέλη υπάρχει ο ίδιος προϋπολογισμός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να εξευρεθούν νέες λύσεις. Είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται κάτι τέτοιο για, ε, ένα 13, το 13ο έτος κατά σειράν. Πώς μπορεί να υπάρξει σωστός ανταγωνισμός. Θα πρέπει να θέσουμε τέλος στις ιστορικές πληρωμές. Θα πρέπει να μας διέπει η αρχή της αλληλεγγύης και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μιλάμε για ίση μεταχείριση Δεν θέλω να ε, φανώ ε, υπερφύαλος. Θεωρώ ότι οι Πολωνοί αγρότες βρίσκονται σε δυσμενή θέση και νιώθουν ότι μένουν απ' έξω. Θα πρέπει να εισακουστεί η φωνή τους. Θα ήθελα να συζητηθεί αυτό εκ νέου και δεν μιλάμε για τις ε, αλλαγές, τις γενικότερες, αλλά για τις ε, μικρές αλλαγές που είχαμε ζητήσει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιους άνισους όρους ανταγωνισμού. Αντιμετωπίσουμε μία πολύ μεγάλη κρίση και εάν δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, τότε θα ε, επεκταθεί αυτή η κρίση θα ήθελα ο Επίτροπος να ξανασκεφτεί ορισμένες από τις προτάσεις και επίσης ο Επίτροπος ε, υπεύθυνος με τα δημοσιονομικά θα πρέπει να ξανασκεφτεί το ζήτημα διότι τα νέα κράτη-μέλη δεν θα δεχτούν τόσο ασαφείς ε, προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ. Χρειαζόμαστε νέες αρχές και αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα δώσω το λόγο σε, τον, σε έναν υπεύθυνο μιας Ιρλανδικής οργάνωσης συντεχνιών. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Από την Οργάνωση Εργατών της Ιρλανδίας λαμβάνω το λόγο. Θα ήθελα για να είμαι σύντομος να επικοινωθώ σε πέντε σύντομα σημεία. Καταρχήν για τη θέση των συνεταιρισμών. Πιστεύουμε ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να τονίσει και να προωθήσει τη θέση των αγροτών σε συνεταιρισμού. Οι συνεταιρισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη πάντοτε δίνουν ε, πολλά ωφέλη στα μέλη τους και στην αγροτική κοινότητα και στον κλάδο γενικότερα. Είναι ένα μοντέλο βιώσιμο και υπάρχει ολοκλήρωση των ε, παραγωγών και της αγοράς ε, και το μοντέλο ε, οδηγεί σε μια ισορροπημένη αλυσίδα διατροφής βελτιώνει τα εισοδήματα των αγροτών και καλύτερο επιχειρηματικό πνεύμα. Κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και η μεταβλητότητα των παγκόσμιων αγορών. οι συνεταιρισμοί παραμένουν ε, η πιο σωστή μορφή οργάνωσης των αγροτών ε, και όχι οι οργανώσεις ε, παραγωγών και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί με την τωρινή ανακοίνωση. Χαιρετίζουμε μέτρα όπως η δημόσια παρέμβαση και η αποθεματοποίηση και είναι κέρια σημασίας το να υπάρχει κάποια προστασία στους γεωργούς κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως ε, η κατάρρευση του τομέα των γαλακτοκομικών το 2008 θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί θα μπορούν να αντιδρούν όταν υπάρχει κάποια διαταραχή στην αγορά με τρόπο αποτελεσματικό. Τρίτο σημείο, για τους νέους αγρότες, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία το 2% της ΚΑΠ να αφορά τους νέους αγρότες, γιατί σε εμά στην Ιρλανδία μόνο το 7% των αγροτών είναι κάτω της ηλικίας των 35 ετών. Για να μπορέσουμε να έχουμε ε, ε, σωστό, ε, σωστή στόχευση θα πρέπει να έχουμε νέο αίμα στη γεωργία. Επίσης μια προτεραιότητα είναι οι βέλτιστες πρακτικές και η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες κατάρτισης των νέων αγροτών ε, σε τομείς όπως ε, τα οικονομικά και η διαχείριση. Τέταρτο σημείο για το πρασίνισμα της ΚΑΠ χρειάζεται μια λεπτομερής ανάλυση για να δούμε ποια είναι η επίπτωση στους αγρότες επακριβώς, τι δυνατότητες ευελιξίας έχουν τα κράτη-μέλη και τι δυνατότητες υπάρχουν για μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική ευθύνη και τις προκλήσεις που τίθενται για τους συνεταιρισμούς. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία της τωρινή πρότασης για το πρασίνισμα της γεωργίας θα μειώσουν την ανταγωνιστικότητά μας στην παγκόσμια γεωργία. Οι άμεσε ενισχύσει θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο περιβαλλοντικέ πτυχέ, αλλά και τη συνεισφορά στην συνοχή στι αγροτικέ περιοχέ, κάτι το οποίο διασφαλίζει το συνεταιριστικό μοντέλο τα τωρινά μέτρα ε, επιβαρύνουν πάρα πολύ ε, ε, τη δραστηριότητά μας μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης και όσον αφορά την καινοτομία, θέλω να πω ότι η ανταγωνιστικότητα είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί και στην Ιρλανδία και σε όλη την κοινότητα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν είδη διατροφής για τον πληθυσμό του πλανήτη που θα είναι 9 δισεκατομμύρια όπως είπαμε το 2050. Η καινοτομία λοιπόν και η έρευνα είναι απαραίτητα για τη γεωργία και ξέρουμε ότι μέχρι τώρα τη χρηματοδότηση σε αυτούς τους τομείς τους έπαιρναν ακαδημαϊκοί φορείς και οι μεγάλες βιομηχανίες που μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τις πολύπλοκες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε όλο τον κλάδο να επωφεληθεί από την καινοτομία και την έρευνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ε, προϊόντα ε, τα οποία θα έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και όχι απλώς πρώτε ύλες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να πω κάτι κι εγώ ως προς την ε, οργάνωση αυτή. Αυτή η συζήτηση σκοπό έχει να βοηθήσει τα τρία θεσμικά όργανα στην εργασία τους για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Στις 7 Νοεμβρίου είχαμε μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση και ήταν η συζήτηση σε επίπεδο ευρωβουλευτών. Σήμερα θα ήταν καλύτερα οι ευρωβουλευτές να ακούσουν τη θέση των εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων. Εάν βεβαίως ε, υπάρχει χρόνος, αφού εκφραστούν όλες οι αγροτικές οργανώσεις, τότε θα ζητήσω από τους ευρωβουλευτές να λάβουν το λόγο. Αλλά επί του παρόντος θα δώσουμε προτεραιότητα στις οργανώσεις των αγροτών. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνέχεια στον κύριο Γκίλιαμ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συμπρόεδρε, ε, κύριες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είμαι αναπληρωτής πρόεδρος, αντιπρόεδρος δηλαδή, της Βρετανικής Οργάνωσης Γεωργών και θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος 47 αγροκτημάτων που εκπροσωπούμε στην Αγγλία και Ουαλία. Καταρχήν θα ήθελα να επαναλάβω το μήνυμα της Ένωσης μας εδώ και καιρό. Τέσσερις αρχές. Πρώτον, απλότης. Να υπάρξει το απλούστερο δυνατό σύστημα στήριξης που να μην απλό μόνο για τους γεωργούς αλλά και για τις κυβερνητικές υπηρεσίες που κάνουν τις πληρωμές γιατί συναντήσαμε τεράστια προβλήματα ως προς αυτό στην Αγγλία. Κοινή πολιτική πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά που να εφαρμόζει πράγματι μια ανταγωνιστική γεωργία που να στηρίζεται στην παραγωγή. Ακούσαμε για τα προβλήματα της ζήτησης περισσότερων φρουτολαχανικών και οι επιστήμονες ακόμη λένε ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή τους κατά 70% μέχρι το 2050 αν θέλουμε να θρέψουμε όλο τον πληθυσμό. Οι Εθνικές Ενώσεις Γεωργών εδώ και καιρό λένε ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή με λιγότερη βλάβη για το περιβάλλον. Πιστεύουμε στην καινοτομία σε πιο σύγχρονες μεθόδους με πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Ήμασταν υπέρ της μεταρρύθμισης Φίσλερ και μέσω των δοκιμών που έγιναν για να οδηγηθεί η γεωργία σε μια κατάσταση που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς. Αν θέλουμε πράγματι να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική γεωργία First of all, πρέπει όντως να δεχτούμε αυτή τη μεταρρύθμιση για να μειωθεί η, γεω... γραφειοκρατία και το κόστος για τα μέλη μας γιατί αυτό θα αυξήσει τις τιμές των τροφίμων μακροπρόθεσμα. Είδαμε από την αξιολόγηση ότι το κόστος αυξάνεται πολύ ιδιαίτερα ως προς το χείριο κρέας και τις όρνηθες, τα πουλερικά. Εμείς δεν είμαστε κατά των βελτίστων πρακτικών υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά θέλουμε η ποιότητα και όχι η ποσότητα να είναι η βάση. Το 75% των γεωργών της Αγγλίας και της Ουαλίας συνυπέγραψαν προτάσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουν μειωθεί κατά 30% τα λοιπάσματα και έχουν φυτευτεί πολλά χιλιόμετρα και μίλια διαχωριστικών θάμνων. Στα Midlands της Αγγλίας με τον υπουργό μας κύριο Jim Pace επισκεφθήκαμε ένα αγρόκτημα όπου η οικογένεια μέσω μιας εθελοντικής φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής του τα τελευταία πέντε χρόνια είχε αυξήσει κατά 40% την παραγωγή της. Αυτό αποδεικνύει ότι το θέμα είναι η ποιότητα. Αυτή τη στιγμή ακούγονται ανησυχίες των γεωργών της Αγγλίας και της Ουαλίας ότι θα χρειαστεί να ανανεώσουν τα εθελοντικά αυτά τους προγράμματα. Θα ήθελα να μας εγγυηθεί ο η Κομισιόν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε οι γεωργοί αυτοί δεν θα τιμωρηθούν, δεν θα ζημιωθούν μέσω των υποχρεωτικών αγραναπάφουσεων. Επίσης μας ανησυχεί ιδιαίτερα το κάπινγκ. Ιδιαίτερα λόγω της γραφειοκρατίας που θα απαιτήσει. Οι Ουαλοί θέλουν μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για να περάσουν στο νέο σύστημα πληρωμών. Για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων οι αλλαγές θα είναι υπερβολικά απότομες και χρειαζόμαστε και εκεί με μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Η Εθνική Ένωση Γεωργών θέλει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις Επαναλαμβάνω λοιπόν το μήνυμα απλότητα, κοινοτικό χαρακτήρας με βάση την αγορά και την παραγωγή. Φοβάμαι ότι αν αυτές οι προτάσεις, ιδιαίτερα τα θέματα του πρασινίσματος εφαρμοστούν, τότε οι Ευρωπαίοι γεωργοί ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Παρακαλώ λοιπόν να στρέψετε την προσοχή σας προς τους κανόνες προς μια βάση αγοράς για να γίνουμε και εμείς πραγματικός οικονομικός τομέας μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα βιολογική παραγωγή. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αναφερόμενοι στα σχόλια του συναδέλφου εξ της Βία Καμπεσίνα, θα ήθελα να σας πω ότι όλοι μπορούμε να οργανώσουμε συζητήσεις, αλλά εσείς ε, ως Πολωνική Προεδρία θα πρέπει να φιλοξενείτε όλους τους φορείς και μα δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είναι σαν να έχετε μία οικογενειακή συνάντηση των παλαιών οικογενειών και της διατροφικής αλυσίδας και δεν ε, προσκαλέσατε ένα ευρύτερο δίκτυο ε, εμπλεκόμενων φορέων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται η ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Βεβαίως οι αγρότες είναι το επίκεντρο της ΚΑΠ και εγώ εκπροσωπώ τον αγροτικό κόσμο και γνωρίζω ότι πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων και θα πρέπει να βρούμε μία κοινωνική συνενετική βάση έτσι ώστε να γίνουν και, για, και εξοικονομήσεις. Επίσης υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς που, που είναι οι ομάδες που αφορούν την ευημερία των ζώων, το περιβάλλον, οι μελισσοκόμοι, δεν τους βλέπω εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω αυτή τη μεγάλη απογοήτευση. Έγινε λόγος για ανταγωνιστικότητα στις συζητήσεις. Έχω την εντύπωση ότι αναπαράγεται ένας μύθος, διότι τη στιγμή που εξαρτώνται από την υποστήριξη όλων οι αγρότες, τότε δεν εκπροσωπούν μία ανταγωνιστική αγορά. Βεβαίως βασιζόμαστε στην υποστήριξη αυτή. Όλοι θέλουμε να υπάρξει μία κοινή αγροτική πολιτική που να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και να διασφαλίζει την εργασία των αγροτών. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, έναν αγώνα τιμών προς τα κάτω για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να έχουμε μια ποιοτική παραγωγή, διαφοροποιημένες αγορές και να μας ενδιαφέρουν οι δίκαιες τιμές εάν θέλουμε να προμηθεύσουμε την αγορά και να εξασφαλίσουμε δίκαιες τιμές στους εργαζόμενους για, και στους αγρότες για να σέβονται και το περιβάλλον. Οι αγρότες οργανικών παραγωγών θέλουν να εργάζονται εδώ και χρόνια για να προστατεύσουν και το περιβάλλον και βεβαίως πρέπει να λάβουν αυτό το πριμ, αυτό το μπόνους. Επίσης πρέπει να διατηρήσουμε την παραγωγικότητα αυτού του τομέα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την παραγωγικότητα, αλλά όχι όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Μιλάμε για φυτοφάρμακα, ενέργεια, φυτοκτόνα, παρασιτοκτόνα μάλλον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έχουμε μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της ενέργειας στο μέλλον. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε λοιπόν από αυτές τις εισαγωγές στο μέλλον. Θα πρέπει οι αγρότες να μπορούν να επενδύσουν σε ένα εκτενές γεωργικό σύστημα με καλύτερη χρήση των πόρων μας και να αλλάξουμε και το όλο σύστημα της αλυσίδας διατροφής για να κάνουμε καλύτερη χρήση των πόρων, να μιλήσουμε για βιοπικιλότητα και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι η βιωσιμότητα είναι, ένα, είναι ο πρώτος πυλώνας, αλλά χρειαζόμαστε και έναν δεύτερο για να προωθήσουμε την διατροφική ασφάλεια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι στο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να λάβουμε μέτρα δυνάμει του Natura 2000, την παραγωγή με οργανικά μέσα, καθώς και να υπάρχει συνεχής έλεγχος των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι ένα σχόλιο. Για δύο εβδομάδες ε, έλεγα σε οργανώσεις Πολωνών ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, αλλά σε 20 χρόνια κατά την επόμενη Πολωνική Προεδρία θα γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση και θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλες τις αγροτικές οργανώσεις, χιλιάδες ανθρώπους που θα παρίστανται. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, Γενικό Γραμματέα. Της Κόπα. Πρόεδρε Σαβίτσκι, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κύριε Επιτρόπε. Συμφωνώ με τους άλλους δύο προέδρους, τον κύριο Ζοντ Λάιτνερ και τον κύριο Μπρούνι. Αυτό δεν θα σας εκπλήξει. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τα θέματα διαδικασίας στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Συμφωνώ επίσης με τη συνάδελφο Γκέλεκ όταν μίλησε για την παλαιά οργάνωση Κόπα Κοζέκα. Συμφωνώ. Ε, είναι ήδη 53 ετών η οργάνωσή μου και εγώ γύρω στα 50, άρα έχει δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπαίνει σε μειονεκτική θέση η κόπα Κοζέκα, γιατί είναι παλαιότερη από άλλες οργανώσεις σε αυτήν την αίθουσα. Η ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ συμφωνεί με τη διαδικασία στην απόφαση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στην κοινή αγροτική πολιτική. Επίση, συμφωνούμε με τι υπηρεσίε τη Επιτροπή και τον Επίτροπο Τσιόλο, ε, που μα είπε ότι υπάρχουν ε, τρεις ε, ε, διαστάσεις στην κοινή αγροτική πολιτική στο μέλλον. Η ασφάλεια των τροφίμων, η επιστηστική ασφάλεια, η ισορροπημένη ανάπτυξη και η εδαφική ανάπτυξη. Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι και επιχειρήματα της Κόπα Κοζέκα και χαιρόμαστε που έχουν ληφθεί υπόψη και τα δικά μας μελήματα. Τι διαφέρει όμως τώρα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Διαφέρει το ότι πρέπει η αλυσίδα των τροφίμων να λειτουργήσει στο μέλλον πολύ καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα. Αντίθετα με κάποιους άλλους ομιλητές που έλαβαν το λόγο, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην εσωτερική αγορά πρέπει να πείσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστιθέμενη αξία την οποία μπορούν να παράσχουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις μας και να έχουμε απόδοση για τις επενδύσεις των αγροτών ανεξάρτητα από τις ε, μεθόδους παραγωγής και το είδος των προϊόντων τους. θα πρέπει να συμβαδίζουμε με τις προτιμήσεις των πολιτών και των καταναλωτών, να ακούμε τι θέλουν να παράγουμε. Εμείς λοιπόν ως Κόπα Κοζέκα και εγώ ως Γενικός Γραμματέας, καλώ όλους τους εμπλεκομένους που έχουν σχέση με τη διατροφική αλυσίδα, κυρίως τις βιομηχανίες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το συνάδελφο από τη Δία Καμπεσίνε, τον κύριο Σομπλάν που έλαβε το λόγο, όλους τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, ε, τον κλάδο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ιδιαίτερα να λάβουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα παλέψουμε για τον τομέα της γεωργίας που θέλουμε να γίνει πιο αποτελεσματικός και να έχει μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη. Η Κόπα Κοζέκα συνεργάζεται με όλους τους φορείς και στόχος μας πρέπει να είναι και τα 13 εκατομμύρια των Ευρωπαίων αγροτών και οι οικογένειές τους θα πρέπει να μπορούν να έχουν επαρκή εισοδήματα από τη γεωργία και να μπορούν ε, να ζουν σε περιοχές που ευημερούν. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει και άλλους παράλληλους στόχους. Όμως αυτός είναι ο πλέον σημαντικός στόχος κατά τη γνώμη μας. Και Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν την ίδια γνώμη. Οι αγρότες και οι οικογένειές τους βρίσκονται πραγματικά στην καρδιά της ΚΑΠ, ανεξάρτητα από το αν θεωρούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι πρόσθετοι στόχοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο των αγροτών από τη Λετωνία, Κλάους Άρμα. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Σαβίτσκι, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκπροσωπώ τη Λετωνία και τις ε, αγροτικές μας οργανώσεις. Άκουσα τον εκπρόσωπο των οργανικών καλλιεργειών θα ήθελα να πω ότι και εγώ εκπροσωπώ τους μελισσοκόμους της Λετωνίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το, την Επιτροπή για το, τα όσα έκαναν για τη μελισσοκομεία στα πλαίσια των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι Λετωνοί αγρότες ε, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Με συγχωρείτε. Ε, εμείς ως Λετονοί αγρότες ε, λαμβάνουμε το, τα χαμηλότερα ποσά ε, άμεσων πληρωμών. Θεωρούμε ότι η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κάνει καλή κατανομή των άμεσων πληρωμών. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στη Λετωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και η ανταγωνιστικότητά μας ε, υποσκάπτεται. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η πρόταση δεν αντικατοπτρίζει αυτά που μας είχατε υποσχεθεί. Το 2008 η Επιτροπή είχε αναφέρει το 2008 και το 2010 ότι θα υπάρχει ίση κατανομή, γι' αυτό και, ε, και έγινε επανακατανομή των άμεσων πληρωμών. Θεωρούμε ότι η αρχή αρχές, ο, ο τρόπος υπολογισμού άμεσων πληρωμών είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος. Θα πρέπει να δείτε ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια που ισχύουν σήμερα και αντικατοπτρίζουν το εργατικό κόστος, ε, το κόστος της γης, τον, ε, του εξοπλισμού, του αγροτικού εξοπλισμού και ούτω καθεξής. Αυτά τα πεπαλαιωμένα στοιχεία δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται. Τα τρία βαλτικά κράτη θα είχαν ε, περισσότερη υποστήριξη εάν είχαμε έναν νέο τρόπο υπολογισμού των άμεσων πληρωμών. Θεωρείται ότι το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλό. Στη χώρα μου, στη Λετωνία για παράδειγμα, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν Υπάρχουν ορισμένες παραγωγές που έχουν χαμηλότερο κόστος από άλλα κράτη-μέλη, αλλά κατά μέσο όρο το κόστος παραγωγής δεν είναι χαμηλότερο από αυτό της Δυτικής Ευρώπης. Οι τελευταίες στατιστικές το, το αποδεικνύουν αυτό. Οι οργανώσεις των αγροτών θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι άμεσων πληρωμών που θα είναι το 80% του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά ε, ε, δεν θα ήταν λογικός ο τρόπος το κόστος μας και οι δαπάνες είναι παρόμοιες με τις δικές σας, γι' αυτό και οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να, είναι, να προσεγγίζουν αυτές της Δυτικής Ευρώπης. Από το 2013 δεν θα είμαστε σε θέση να καταβάλουμε άμεσες πληρωμές στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης στη Λετωνία για να μην στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά δεν καταλαβαίνουμε την ε, συλλογιστική σας και τη λογική που διέπει αυτή τη νέα πρόταση. Επίσης, πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή δεν είναι ισορροπημένη. Πριν συνοψίσω, θα ήθελα να μιλήσω για τους νέους αγρότες. Χρειάζονται υποστήριξη, αυτό είναι, θα πρέπει να είναι ένα δεσμευτικό βήμα για όλες τις παραγωγές, για τους νέους γεωργούς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους ε, αγρότες στη Λετωνία, διότι κινδυνεύει να εκλείψει το είδος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η Φινλανδία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Λέγομαι Σίμωτι Άινεν και είμαι διευθυντής του Γραφείου Βρυξελών της ΕΝΤΕΑ, δηλαδή των Φιλανδών Δασοκόμων και Γεωργών. Ευχαριστώ όλους όσους, όλους όσοι συμμετέσχουν εδώ στην εκδήλωση που είναι τόσο σημαντική γιατί συζητάει το μέλλον της ΚΑΠ. Οι προτάσεις της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ περιέχουν στοιχεία πολύ θετικά για μας και που θα τα υποστηρίξουμε. Οι Φιλανδοί Γεωργοί υποστηρίζουν τους στόχους που εκφράζει η Κομισιόν για να συνεχιστεί βιώσιμη αγροτική παραγωγή σε ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει όμως και οι διαφορές να γίνουν σεβαστές γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η ΚΑΠ να είναι πράγματι κοινή. Η στόχη της Κομισιόν δηλαδή η ενδυνάμωση της θέσης των παραγωγών είναι κάτι το τελείως ουσι... ουσιώδες. Επίσης οι στηρίξεις με βάση την παραγωγή είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για τη Φιλανδία όπου είναι πολύ ψηλό το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Δυστυχώς από την άλλη μεριά οι προτάσεις αυτές εμπεριέχουν και ορισμένες αδικίες που θα έπρεπε να διορθωθούν. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ακόμη πολλή δουλειά για να το καταφέρουν και θα χρειαστούν και άλλες συζητήσεις σαν Στην πρότασή της η Κομισιόν δεν προσέχει επαρκώς το θέμα της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής για την εγγύηση των αγροτικών εισοδημάτων και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Παραδείγματο χάρη, ό,τι λέγεται για το πρασίνισμα της γεωργίας δεν γίνεται δεκτό από τους Φιλανδού γεωργούς οι οποίοι ήδη σε εθελοντική βάση έχουν λάβει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και αυτά που προτείνει η Κομισιόν για το λεγόμενο πρασίνισμα της ΚΑΠ θα μεταφράζονταν σε περισσότερη γραφειοκρατία και υψηλότερο κόστος της παραγωγής. Η πρόταση παραδείγματο χάρη που αφορά τις τρεις καλλιέργειες της διαθέσιμες γέες είναι κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Επίσης οι λεγόμενες επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος είναι κάτι πολύ αμφίβολο για μας. Δεν συμβαδίζει με την απαιτούμενη αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας. Ο ορισμός αυτών των επιφανειών είναι επίσης ασαφής. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο Τσόλος το εξής. Ποιες είναι οι επιφάνειες που μπορούν να θεωρηθούν ως οικολογικού ενδιαφέροντος, όλες. Και πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταλήξουν όλα αυτά σε περισσότερο γραφειοκρατικό και διοικητικό άχθος για τους παραγωγούς. Η οργάνωσή μου θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει ότι πραγματοποίηση των προτάσεων αυτών της Κομισιόν για τη μελλοντική ΚΑΠ εξαρτάται βασικά από τις αποφάσεις χρηματοδότησης που θα ληφθούν και μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία πληροφορία για τη χρηματοδότηση που θα επέτρεπε την εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί μια ισχυρή ΚΑΠ αλλά με τρόπο ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και τώρα η εκπρόσωπος της Ισπανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την Αζάχα, μια ισπανική οργάνωση που έχει πάνω από 5.000 μέλη. Ως παρατηρητής συμμετέχω εδώ στη συζήτηση Άλλοι όμως θεωρούνται πιο σημαντικά μέλη φαίνεται και δεν είναι παρατηρητές αλλά πλήρη μέλη. Ερωτώ παρόλα αυτά τον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, η πρότασή σας έχει πολλά θετικά στοιχεία όπως διαφοροποιημένη μεταχείριση ανατομέα. Αλλά και η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι κάτι το θετικό. Πρόκειται για νέα μέτρα που ενδιαφέρουν πολύ τους νέους αγρότες. Όλα αυτά είναι θετικά, επαναλαμβάνω. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες ελλείψεις και ορισμένες απορίες μας τίθενται, παραδείγματος χάρη. Το δικαίωμα ορισμένων χωρών, όπως η δική μου, όπου υπάρχουν πολύ διαφορετικές επιφάνειες και ετερογένεια, είναι απαραίτητο να κάνει τη μετάβαση στα νέα μέτρα με μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο, μέχρι το 21. Αυτό το 40% που προβλέπετε αρχικά δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλό, 20% να βάλετε στην αρχή. Υπάρχουν πολλές σημαντικές ιδέες που πρέπει όμως να τις συμπληρώσετε γιατί ήδη ακούγονται πολλά. Οι επιλεγμένες επιφάνειες δεν είναι κάτι που ορίζεται συγκεκριμένα. Τα βοσκοτόπια τι θα γίνουν. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και θα πρέπει η Κομισιόν το συντομότερο δυνατόν να μιλήσει για μεταφορά δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα ε, επιμέρους θέματα όπως ας πούμε η συγχώνευση, υπάρχει η επίμορτος αγροληψία και άλλα θέματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει διάκριση του 80% των αγροτών που λαμβάνουν κάτω από 5.000 ευρώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο αυτός ο αγρότης είναι ενεργός. Εντάξει, να απλουστεύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να ε, σταθούμε και να δράσουμε κατά των μικρών γεωργών. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες αγρότες και εσείς δημιουργείτε ε, μεγαλύτερη γραφειοκρατία και περισσότερους ε, ελέγχους ως προς το, την ε, πράσινη γεωργία. Μερικοί έλαβαν ήδη τις επιδοτήσεις, εγώ όμως όχι. Όσο και να γίνεται λόγος για αυτή την πράσινη καταβολή, δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται στον πρώτο πυλώνα. Θα έπρεπε να βρίσκεται στον δεύτερο, έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή με την αιρεσιμότητα. Όταν μιλάμε για οικολογική γεωργία, θα πρέπει να την χάνει της ίδιας μεταχείρισης, όπως άλλοι παραγωγικοί τομείς. Αυτό το μήνυμά σας για τους νέους γεωργούς δεν αρκεί οι νέοι γεωργοί ζητούν αλλαγές στη λειτουργία της διατροφικής αλυσίδας ή του ανταγωνισμού. Βεβαίως, ε, συνεργάζεστε και με τον Επίτροπο Αλμούνια και με άλλους συναδέλφους, αλλά θα πρέπει να έχετε σωστές τιμές που να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Γιατί πολλές από τις προτάσεις σας για την διαχείριση του κινδύνου δεν, είναι, δεν θα έχουν αντίκρισμα. Και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερο. Και αυτό απασχολεί και τους νέους γεωργούς. Ευχαριστώ πολύ. Η Εστονία έχει το λόγο. Ο, η εκπρόσωπος της Εστονίας. Ευχαριστώ. Ως εκπρόσωπος ε, των γεωργικών οργανώσεων τη Εσθονία, θέλω και εγώ να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα ή τις συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού που ε, επίσης εντοπίζουμε στην πρόταση της Επιτροπής. Η Εσθονία όπως και άλλες χώρες της επιτροπη η εσθονια οπως και αλλες χωρε της βαλτικη δεν συμφωνεί με την ε, εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων. Δεν γίνεται με το σωστό ρυθμό και δεν παρέχονται επαρκείς όροι ανταγωνιστικότητας για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, άρα χρειαζόμαστε μια μεταβατική περίοδο μιας γενιάς και αυτό δεν συνάδει προς τη βιωσιμότητα της γεωργίας μας ε, και την διατροφική ασφάλεια. Παράλληλα υπάρχει μετακίνηση των ε, πολιτών από τις αγροτικές περιοχές της πόλης και όχι μόνο στις πόλεις αλλά και σε άλλες χώρες. Και όπως είπε συνάδελφος από την Λετωνία, λειτουργούμε μέσα σε μια κοινή αγορά και έχουμε τους ίδιους στόχους και ίδιες απαιτήσεις. Και η παραγωγή μας δεν είναι πιο φθηνή από ότι στο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα θέλαμε το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων σε όλες τις χώρες να είναι το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη περίοδο και θα θέλαμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία που μας δίνεται και να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τις τρευλώσεις ανταγωνισμού που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και όλα τα άλλα μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλοι ο Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βόντι Σαφή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά μέλα, μέλη, ε, η μεταρρύθμιση αυτή είναι η ύψη της σημασίας για τους Πολωνούς αγρότες και αυτό που λέγεται συνάδει με αυτό που είπαν και άλλοι εκπρόσωποι από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Προσπαθούμε να πείσουμε έτσι προσπαθήσαμε να πείσουμε τους Πολωνούς ε, πολίτες να δεχτούν την προσχώρηση της χώρας. Είχαν δοθεί πολλές υποσχέσεις και είχε υποθεί ότι η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι το 2013. Τώρα όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παρατείνει την μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μιλάμε για διαφοροποίηση της ε, παραγωγής με βάση την ε, διαφοροποίηση των πληρωμών. Αυτό κάνει η μεταρρύθμισή σας. Το ίδιο ισχύει στα βαλτικά κράτη, στην τσεχική δημοκρατία και στην Πολωνία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει μια σωστή πλατφόρμα και ίσους όρους πρόσβασης. Οι συνάδελφοι από την Πολωνία και τα άλλα, άλλα κράτη-μέλη που εκπροσωπούν τα 12 νέα κράτη-μέλη λένε ακριβώς ότι υπάρχουν ανισότητες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε ίσους όρους πρόσβασης. Το κόστος είναι το ίδιο, οι δαπάνες μας είναι οι ίδιες, γι' αυτό χρειαζόμαστε ίση μεταχείριση, γιατί μόνο έτσι τα μετασοσιαλιστικά αυτά καθεστώτα θα γίνουν ανταγωνιστικά. Θεωρήσαμε ότι τα επτά χρόνια θα ήταν αρκετά και μας προτείνατε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Δεν θέλουμε να αποσπάσουμε χρήματα από Γάλλους ή Γερμανούς αγρότες. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες με όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει η μεν να στραφούμε κατά τον δε. Δεν πρέπει να θεωρηθούμε ανταγωνιστές γιατί προερχόμαστε από την Πολωνία ή την Εσθονία. Πιστεύω ότι η αρχή του πρασινίσματος και αυτό το 7% είναι κάτι για να μας αποσπάσει την προσοχή από άλλα στοιχεία. Διότι οι αγροτικές οργανώσεις και ενώσεις λένε ακριβώς αυτό, ότι αυτό ενυπάρχει για να μας αποσπάσει την προσοχή από την ουσία, δηλαδή από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την ΚΑΠ και εγώ νιώθω υπεύθυνος και λογοδοτώ σε όλους τους αγρότες, διότι ήμουνα μεταξύ εκείνων που προσπάθησα να πείσω τους Πολωνούς αγρότες ότι θα ήταν ευεργετικό να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι μας μεταχειρίζεστε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ένα άλλο θέμα είναι οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί. Ο Υπουργός μας ε, λέει ότι αυτό το ζήτημα είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μεμονωμένων κρατών. Ως προς τις, ε, τους συνεταιρισμούς, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η κάθε συντεχνία απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζόμενους. Και στην ε, Πολωνία πολλοί προσπαθούν να φύγουν από τους συνεταιρισμούς. Γι' αυτό θέλουμε να μας βοηθήσετε για να πείσουμε τις πολωνικές αρχές ότι οι συνεταιρισμοί οργανώνουν καλύτερα την αγορά και ότι υπάρχουν ευεργετικοί ε, μηχανισμοί. Ο Υπουργός Σαββίτσκι μας υποστηρίζει, αλλά η υποστήριξή του δεν επαρκεί. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχέδιο μεταρρύθμισης θα πρέπει να αλλάξει και περιμένουμε τις νέες σας προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ένας αυστριακός εκπρόσωπος. Σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής κύριε Ντακάστρο, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω εν συντομία το λόγο εδώ και να μιλήσω εκ μέρους ε, του, του Γεωργικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας. Γεωργ Κάμερ είναι το όνομά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις της Επιτροπής που μας έχετε υποβάλει που περιλαμβάνουν πολλές θετικές πτυχές. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τονίσουμε τις θετικές πτυχές, γιατί πότε δεν έχουμε το χρόνο να τονίσουμε τα θετικά. Πάντοτε πρέπει να κάνουμε παρατηρήσεις για αυτά στα οποία έχουμε αντιρρήσεις. είναι σημαντικό να τονίσουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, όπω είπαν και προηγούμενοι ομιλητέ, και τι παράλληλε διαδικασίε όσον αφορά τον προπολογισμό θα πρέπει να προβλέπονται και για τη γεωργία επαρκή σπόροι για να μπορέσουμε να φροντίσουμε το μέλλον της ε, κοινή αγροτικής ε, πολιτικής. Ε, παράλληλα υπάρχει η πτυχή του περιβάλλοντος που λαμβάνεται υπόψη το νέο προϋπολογισμό και εδώ υπάρχουν μέτρα τα οποία εν μέρη ήδη λαμβάνουν χώρα σε θελοντική βάση πολλές φορές και θα θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα με ευέλικτο τρόπο να βρεθεί μια λύση αποφεύγοντας το υπερβολικό κόστος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αναφέρθηκε η βιολογική γεωργία και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Θέλουμε να υπάρχει μια παρόμοια μεταχείριση ε, για τις διάφορες μορφές γεωργίας. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ε, θα ήθελα να μιλήσω για την κατανομή στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, γιατί υπάρχουν χώρες που για ιστορικούς λόγους εφαρμόζουν το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων και θα πρέπει να τους αφήσουμε επαρκή ευελιξία για να προσαρμοστούν ε, στον, ε, στα νέα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των περιφερειών τους και να μην υπάρχουν ε, μεγάλες διαταραχές στα κράτη-μέλη λόγω ε, των ε, νέων των παραγόντων που υπάρχουν στις προτάσεις μεταρρύθμισης της Επιτροπής. Και επίσης μας ενδιαφέρει να τονίζουμε το ρόλο των ενεργών αγροτών η διαχείριση της αγοράς ε, είναι ένα σημαντικό τομέας και εδώ θα πρέπει να, να τονίσουμε και να εξετάσουμε όλες τις επιπτώσεις ε, ε, των μέτρων που λαμβάνονται είτε για την κατάργηση κάποιων μέτρων στήριξης είτε για την παράταση κάποιων οργανώσεων αγοράς. Ευχαριστώ και την Κόπα Κοζέκα για όσα μας είπε και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η κοινή αγροτική πολιτική λειτουργεί σωστά για τους αγρότες όταν θέτει κίνητρα που να ε, είναι καλά και για τις οργανώσεις παραγωγών και για τις ε, οργανώσεις νέων αγροτών. Οι νέοι αγρότες είναι πολλοί στην Αυστρία και ελπίζω και στο μέλλον να είναι πολλοί και να πολλαπλασιάζονται. Άλλο ένα σημείο για την κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική προσπαθεί να αποφύγει στρεβλώσεις και προς το εσωτερικό αλλά και προς τα έξω και νομίζω ότι στο μέλλον θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών γιατί η αγροτική πολιτική θα μπει στο μικροσκόπιο και θα πρέπει να βρούμε την αγροτική πολιτική που θα ταιριάζει με τους όρους της διεθνούς κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δίνουμε τώρα το λόγο στον πρόεδρο του, του Γεωργικού Επιμελητηρίου και στην πρόεδρο της ΚΟΠΑ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση αυτής της συζήτησης και για όσα μπορέσαμε να μάθουμε κατά αυτήν. Οι γεωργοί που παρίστανται εδώ ανεξάρτητα από το αν εκπροσωπούν τα παλαιά 15 μέλη ή τις νεότερες χώρες, έχουν αντιδράσει με τρόπο που δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιητικέ πλήρως οι προτάσεις αυτές. Διότι η Γεωργία ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία προέρχονται δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτές τις προτάσεις. Κύριε οποια προερχονται δεν ειναι ευχαριστημενη με αυτες τις προτασεις κυριε επιτροπε οι 700 σελίδες της πρότασης τις εκτιμούμε ιδιαίτερα, αλλά θα θέλαμε μια πλούστερη μεταρρύθμιση. 20-30 σελίδες. Γιατί όλες αυτές οι σελίδες που καταλήγουν στο ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι πολύ δυσνόητη και για τους αγρότες και για τις οργανώσεις τους αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες προκλήσεις και καινούργιες προκλήσεις. Αντί λοιπόν να παρατείνεται ορισμένα απαρχαιωμένα μέτρα θα έπρεπε μάλλον να οργανώσετε την Ευρωπαϊκή Γεωργία με τρόπο ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική διεθνώς και πιο ικανοποιητική για τους καταναλωτές και καταναλώτριες. Εμείς δεν συμφωνούμε με μια ΚΑΠ που να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, να αυξάνει το κόστος και να είναι και δυσνόητη η καινούργια ΚΑΠ δεν διασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερη παραγωγή. Είναι πάλι αυτά που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Διατηρείται το status quo πάση θυσία. Οι προκλήσεις υπάρχουν ήδη, είναι παρούσες. Και η εισαγωγή νέων ε, στοιχείων όπως το πρασίνισμα και το 7% set site δεν είναι αποδεκτές προτάσεις. Δεν ξέρουμε ε, γιατί γίνονται αυτές οι προτάσεις, σε τι στοχεύουν. Τι είναι ενεργός παραγωγός που λέτε. Δεν το καθορίζετε σαφώς. και απλώς προσπαθείτε να κρύψετε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην Ήπεθρο. Η αρχή της μεταφοράς κονδυλίων φαίνεται είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει παραπάνω και από την ίδια την γεωργική πολιτική. Η στόχοι της μεταρρύθμισης γίνονται κατανοητοί από όλους, αλλά οι μέθοδοι που επιλέξατε για να τους εφαρμόσετε, για να τους επιτύχετε, απορρίπτονται εδώ όπως είδατε, όπως ακούσατε από τους παρόντες γεωργούς. Το 30% πρασίνισμα τι σημαίνει, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς η παραγωγή οποροκυπευτικών ας πούμε γιατί μπορεί αυτά τα μέτρα τελικά να καταλήξουν σε λιγότερη ανταγωνιστικότητα διεθνώς. Ο Λυκίσκος ιδιαίτερα είναι προβληματικός. Δεν θα μπορέσουν καν να επιβιώσουν στη διεθνή αγορά η παραγωγή του με αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Επίτροπε να καταλάβετε ότι η Κομισιόν δεν χρειάζεται να γράφει όλο και περισσότερες σελίδες αλλά αντίθετα να προτείνει απλούστερα μέτρα και δράση μάλλον αντί για λόγια. Είναι δύσκολο βέβαια να απλοποιηθεί το σύστημα, αλλά πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να τελειοποιηθεί το σύστημα, συμφωνούμε, αλλά νομίζω είναι λάθος ο δρόμος. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο εκπρόσωπος των Ιταλών Γεωργών της Ομοσπονδίας Ιταλών Γεωργών. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Τους κυρίους Σαβίνσκι, Ντεκάστρο, τον ε, Επίτροπο Τσόλος. Έχει μεγάλη σημασία το ότι μπορούμε να εκφραστούμε. Είμαι ο Ρομπέρτο Καβάτσο και εκπροσωπώ την Ομοσπονδία Ιταλικών Συνεταιρισμών. Ναι. Δεν θα είμαι διεξοδικός, απλώς θα ε, μιλήσω για ορισμένες πτυχές της ε, πρότασής σας, διότι περισσότερες γεωργικές οργανώσεις προσχώρησαν σε αυτές τις θέσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Εμείς Θέλουμε απλώς να τονίσουμε ορισμένα στοιχεία. Η ΚΑΠ θα πρέπει να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία αυτού του τομέα, αλλά να λάβει υπόψη και την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ποιοτικών τροφίμων. Θα πρέπει η γεωργία να είναι πιο βιώσιμη και να προωθήσει αυτούς τους στόχους με βάση τα δίκαια εισοδήματα για όλους. Η κατανομή των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να είναι δίκαιη. Και ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, χρειάζεται βαθμιαία καταβολή. Η παράμετρος της επιφάνειας όμως δεν είναι σωστή για την κατανομή των πόρων γιατί η βάση δεδομένων των πληρωμών θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για να λάβουμε υπόψη τους αμπελώνες και τους οπορώνες που δεν ε, ε, λαμβάνονται υπόψη. Πρόκειται για 3 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία δεν λήφθησαν υπόψη. Γενικότερα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν και άλλοι παράμετροι το, η προσθεμένη αξία της παραγωγής και η αυτόνομη εργασία, η ανεξάρτητη εργασία που προωθείται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η αποκλειστική χρήση της ε, έκτασης δεν είναι το σωστό κριτήριο και πιστεύουμε ότι διοικητικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ενιαία. Νομίζω λοιπόν ότι ο αρχηγός εκμετάλλευσης θα πρέπει να ορίζεται σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να υπάρχει και μία ευρωπαϊκή υπόδειξη, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν. Ως προς τις άμεσες πληρωμές θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφορούν τους επαγγελματίες γιατί απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Ως προς το greening και την αύξηση των πόρων συμμεριζόμαστε αυτό το κριτήριο. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ κόστους και δεσμεύσεων προς τους γεωργούς. Και εδώ μιλάμε για ένα 30% των άμεσων πληρωμών. Θα πρέπει να έχουμε ένα φάσμα μετρήσεων το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί. Αν λάβουμε υπόψη τη γεωργία στην κάθε χώρα. Τα ποσά για το πρασίνισμα θα πρέπει να καταβάλλονται και να δαπανώνται από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε επίσης τον υδροφόρο ορίζοντα και τις εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να μιλάμε για ομαδοποίηση της παραγωγής, καθώς και διαχείριση κινδύνων και ασφάλεια εισοδημάτων. Τέτοια μέτρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά γιατί θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διάρθρωση και να προωθείται η εμπορία με καλύτερη οργάνωση. έτσι ώστε να υπάρχει και μείωση γραφειοκρατίας. Επίσης, ως προς τα ασφαλιστικά συστήματα θα πρέπει να υπάρχει μικρότερος φόρτος για να υπάρχει και ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Ως προς την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να προωθούν απροφηθούν απλουστεύσεις, ιδιαίτερα για τους μικροπαραγωγούς και μιλάμε για μεγαλύτερες ποσοστίες αναλογίες καλλιεργειών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική και οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία πολυετή βάση υπολογισμού γιατί χρειάζονται πιο ευέλικτοι μηχανισμοί υπολογισμών και πληρωμών για να φτάσουμε στη... στους στόχους μας. Εμείς θέλουμε να βελτιωθούν αυτές οι προτάσεις οι οποίες αποτελούν μια καλή βάση, ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς, γιατί δεν υπάρχει μέλλον για κανέναν μας αν δεν υπάρχουν οι νέοι γεωργοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μια Ιρλανδική οργάνωση γεωργών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το θέμα που είναι βασικό για την Ιρλανδία και για τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική μετά το 2013. Από την αρχή τη ΕΚΑΠ έχει περάσει από πολλέ μεταρρυθμίσει, προσπαθεί να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των Ευρωπαίων καταναλωτών για ποιότητα και για επαρκή ποσότητα τροφίμων ε, θέλουμε να υπάρχει περιβαλλοντική ισορροπία, εδαφική συνοχή και ανταγωνιστικότητα στη Γεωργία μετά το 2013. Συμφωνούμε με τους στόχους αυτούς και συμφωνούν ε, οι αγρότες με τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ε, θέλουμε οι αγρότες να παράγουν ε, καλής ποιότητας τρόφιμα και να φροντίζουν και για το κλίμα και για την ευημερία των ζώων. Παράλληλα η ΚΑΠ δίνει υποστήριξη για τη συνέχιση του οικογενειακού αγροκτήματος και για την ε, παραγωγή μικρής κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά ανησυχώ, διότι οι προτάσεις της Επιτροπής όσοι έχουν αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε μήπως τυχόν υπονομεύουν τους ενεργούς παραγωγούς και μήπως υπησέρχονται στις αποφάσεις των γεωργών και μειωθεί τελικά η ικανότητα της Ιρλανδικής Γεωργίας να συνεισφέρει στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Φοβούμαι ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις για διασφάλιση επιστηστικής ε, ασφάλεια ε, στην Ευρώπη. Η για πληρωμή αναεκτάριο μέχρι το 2019 ανησυχεί πάρα πολύ τους Ιρλανδούς αγρότες. Σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης οι αλλαγές θα δημιουργήσουν τεράστια ταραχή σε μια δύσκολη περίοδο και θα υπονομευθούν βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι μια πολύ απλουστευτική προσέγγιση και δεν λαμβάνει υπόψη τις βασικές διαφορές στην παραγωγική ικανότητα ε, ε, των διαφόρων περιοχών στην Ιρλανδία. Επίση, θα μειωθούν κατά πολύ οι δυνατότητε παραγωγή των Ιρλανδών αγροτών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ευελιξία για να εφαρμόσουν ένα σύστημα ενισχύσεων που θα υποστηρίζει την παραγωγή, θα διασφαλίζει τι βιώσιμε αγροτικέ επιχειρήσει ε, και τα βιώσιμα επιχειρηματικά ε, συστήματα. Η πρόταση για ένα καταποκοπή ποσό μέχρι το 2019 με έτος αναφοράς από το 2014 και μετά δημιουργεί διαταραχές στην αγορά και θα επηρεάσει τις ε, αποφάσεις των αγροτών. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το εξετάσουμε εις βάθος. Η Ιρλανδία χρειάζεται μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο μετά το 2019 για να υπάρξει η εθνική ανακατανομή. Οι προτάσεις της Επιτροπής για το πρασίνισμα, το greening, θα επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσει ε, στους αγρότες. Τα υφιστάμενα μέτρα ε, πολλαπλής συμμόρφωσης ε, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν από όλους ε, τους εργαζομένους περιλαμβάνουν ε, πολλά μέτρα για την πράσινη ανάπτυξη και τα μέτρα για το πρασινίσμα θα πρέπει να αναθεωρηθούν τόσο ώστε ε, να ενταχθούν στις τρέχουσες λειτουργίες των αγροτών και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν για το περιβάλλον στα διάφορα κράτη-μέλη. Και για ε, την μεταβίβαση του 30% της χρηματοδότησης επίσης πρέπει να επανεξετάσουμε τα μέτρα. Η Ιρλανδία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε πολλά προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου και αναγνωρίζουμε το ρόλο που παίζουν αυτά τα προγράμματα για τη συνέχιση της γεωργίας σε μειονεκτικές περιοχές και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα επίσης είναι σημαντικά. Η μελλοντική χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των διαφόρων περιοχών στην στην παραγωγή στο παρελθόν και θα πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη ευελιξία να εφαρμόζουν μέτρα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον αγροτικό του πληθυσμό και την γεωργική του δομή. Το να παραμείνουν ε, τα υφιστάμενα μέτρα για ε, ε, κρίσει και μέτρα κατεπήγοντα χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικό θέμα σε εποχές κρίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την μεταβλητότητα των τιμών. Όμω θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η πρόταση. Χρειάζεται χρηματοδότηση να βρεθεί χρηματοδότηση για πρόσθετα μέτρα σε εποχές κρίσης, ώστε να έχουν πραγματικό νόημα αυτά τα μέτρα και θα πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα κινητοποιούνται αυτά τα μέτρα. Ε, ανέφερε τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν τους αγρότες στην Ιρλανδία. Όσο προχωρεί η συζήτηση για την ΚΑΠ, πρέπει να πούμε ότι ε, υποστηρίζουμε ε, μια ισχυρή ΚΑΠ στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα, ούτως ώστε να έχουμε επισητιστική ασφάλεια. Και θέλουμε να παραμείνει το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλέ φορές έχουν αλλάξει οι συνθήκες στη Γεωργία και έχουμε προσαρμοστεί και μπορούμε και στο μέλλον να προσαρμοστούμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε ε, σε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Λιθουανίας, των Λιθουανών αγροτών. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ο οργανωτές αυτής της συνάντησης εκπροσωπώ το αγροτικό επιμελητήριο της Λιθουανίας Γιορτάζουμε το 85ο έτος της ε, ύπαρξής μας και είμαστε μέλη της Κόπα Κόζα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Πολωνίας ε, και της, ε, της Πολωνίας, Λετωνίας και της Εσθονίας. Ο εκπρόσωπος των νέων γεωργών είπε ότι θα πρέπει να έχει μια σταθερή βάση η ΚΑΠ. Μιλάμε για αρχές δικαιοσύνης, δημοκρατίας και κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς ε, το λόγο οι τρεις βαλτικές χώρες λαμβάνουν τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές. Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, αυτό ήταν κατανοητό, έτσι είχαν οι διαπραγματεύσεις, αλλά τώρα συνεχίζεται αυτή η βάση, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Ε, γιατί έγινε αυτό, γιατί βρισκόμασταν υποκατοχή 50 χρόνια, γιατί θεωρείτε ότι οι χώρες μας έχουν μικρό μέγεθος. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Όσον αφορά τις απαιτήσει. Οι αρχηγοί εκμετάλλευσης πληρούν τα κριτήρια πολύ καλύτερα από ε, τα παλαιά κράτη-μέλη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο το πρασίνισμα αυτό σημαίνει μείωση του όγκου παραγωγής στην πραγματικότητα, ναι ή όχι. θα πρέπει να παράγουμε και να χορηγούμε τρόφιμα όσον αφορά το πάγωμα γεών, μιλάμε για ένα 7%. Μα πρόκειται για έγκλημα. Πρέπει να δουλεύουμε τη γη και όχι να κάνουμε το αντίθετο. Σήμερα χάνουμε γέες για άλλους λόγους εξαιτίας της αστιφιλίας και μάλλον της ε, ανάπτυξης των μεγάλων πόλεων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να θέσουμε όρους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι για όλους. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ολλανδίας. Ή την εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεκάστρο, Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που μας επιτρέπετε να λάβουμε εδώ το λόγο και θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος των εκπροσώπων των παραγωγών σακχαροτεύτλων στην Ολλανδία. Εκπροσωπούμε το σύνολο των παραγωγών σακχαροτεύτλων και ζάχαρης στην Ολλανδία. Ο τομεύς της ζαχάρεως φαίνεται ότι έχει παραγνωριστεί εδώ στη συζήτηση, έχει αγνοηθεί. Έγινε λόγος για πρασίνισμα, για δεύτερο πυλώνα, για διαφορετική κατανομή των πληρωμών, αλλά η πρόταση της Κομισιόν για τον τομέα μας δεν λέει τίποτα. Φαίνεται ότι τα πρόσθετα μέτρα θα αφορούν μόνο τον τομέα της ζάχαρης. Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι η τωρινή οργάνωση της αγοράς λαμβάνει υπόψη της και τη ζάχαρη, αλλά εδώ μιλάμε για τον προϋπολογισμό των προτάσεων Πράγματι την προηγούμενη περίοδο διαπιστώσαμε μείωση του τομέα στην αγορά, του ρόλου του στην αγορά. Δεν είναι όμως... Δεν οφείλεται όμως αυτό στην απελευθέρωση της αγοράς όπως υπόθηκε, αλλά των μέτρων, είναι αποτέλεσμα των μέτρων που λάβα, λήφθηκαν από την Κομισιόν. Αυτό το ξέρει ως προς τη ρύθμιση των αγορών. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί λοιπόν θα έχουν τη στήριξη που χρειάζονται όπως, την είχε, όπως το είχε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την εξέταση του θέματος της ζάχαρης. Οι προτάσεις του πρασινίσματος ακούγονται εδώ και πολλά χρόνια αλλά εμείς δεν βλέπουμε τι μας αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα. τώρα. Ο επόμενος εκπρόσωπος. Σας χαιρετώ ε, και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Κονράδο ο Ομιλώ ως πρόεδρος του ELO με ένα εκατομμύριο μέλη. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πρέπει να εξασφαλίσει, να προωθήσει την διατροφική ασφάλεια και την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει σωστή ε, διαχείριση των γεών για να φτάσουμε στη βιοπικιλότητα και να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές στην ε, καλλιέργεια των γεών και για να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους. Εμείς μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη μεταρρύθμιση όπως και την προγενέστερη. Υπάρχουν όμως ε, τρία σημεία που δεν είναι καθόλου δελεαστικά. Μιλάμε για την περιπλοκότητα της, της πολυστρωματικής στοχοθέτησης του πυλώνα 1 που είπε ο κύριος Σοτσόλος ότι ελέγχεται εύκολα. Δεν το συμμεριζόμαστε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι ένα περίπλοκο σχήμα και σημαίνει μείωση των ελευθεριών του παραγωγού που είχε προωθήσει η προηγούμενη μεταρρύθμιση διότι τα δύο τρίτα των άμεσων πληρωμών αφορούν μια ε, εκούσια, εθελούσια βάση πέρα από τον πληθωρισμό και υπόθηκε ότι το πρασίνισμα δεν θα αφορά συμβάσεις ε, υπέρ των τροφίμων και του περιβάλλοντος έτσι ώστε να καταβληθεί το τίμημα δύο φορές τους ε, γεωργούς δυνάμει του πυλώνα 1 και 2 με βάση τις βιώσιμες πρακτικές. Όταν μιλάμε για ενεργό αγρότη μπορεί να είναι σκόπιμο να υπάρχει αυτός ο ορισμός όταν μιλάμε για γήπεδα γκολφ. Mm. Αλλά ίσως αποκλείουμε μεγάλες οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, διαφοροποιημένες καλλιέργειες, καθώς και ε, διαχειριστές υδάτινων πόρων. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για ένα 5% κατόφλι το οποίο είναι εφιαλτικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις φορολογικές αρχές και επίσης είμαστε κατά του κάπιν, δεχόμαστε το 25% πληρωμών δυνάμει του πυλών 2, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ορισμένα κράτη-μέλη μπορούν να σταθούν σε ένα 10% άμεσων πληρωμών δύναμη του πυλώνα 2. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τα μέτρα πρασινίσματος θα είναι αποδοτικά με βάση την ε, κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχουν περιβαλλοντικά ευεργετήματα. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει το κόστος καλλιέργειας εξαιτίας του πρασινίσματος, θα αυξήσει τις τιμές της αγοράς, αλλά δεν θα αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος. Η Το παραγωγικό δυναμικό θα μειωθεί ιδιαίτερα για αρρώσιμες γεές και επίσης θα κινηθούμε σε ένα ενοποιημένο δίκτυο για, ο οποίος θα κινείται στις λιγότερο παραγωγικές γέες και αν υπάρχει χαμηλότερη προμήθεια θα υπάρχουν και χαμηλότερες εξαγωγές και συνεπώς η Ευρώπη δεν θα συνεισφέρει τόσο πολύ στο να θρέψουμε τον κόσμο. Άρα θα μειωθεί η διάδραση αυτή και θα μειωθούν και τα εισοδήματα ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ε, εισαγωγές προϊόντων. Τα κίνητρα είναι το καλύτερο μέσο παραγωγής δημοσίων αγαθών και θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους γεωργούς έτσι ώστε η γεωργία να γίνει βιώσιμη όπως ορίζουν οι εκθέσεις Lion και Des. Θεωρούμε ότι η έκθεση Καπούλα Σάντος επίσης θα τονίσει την πτυχή των κινήτρων και όπως προανέφερε ο Επίτροπος Τσόλος δεν έχει λήξει η δημόσια συζήτηση και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι φτάνουμε στο τέλος των ομιλητών μας θα έχουμε δύο, έναν και έναν ομιλητές. Από την αριστερά, το, τα μεσαία έδρανα και τα δεξιά. Εγώ ονομάζομαι Βάιντεσεύσκι και συμμετέχω στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ε, εκπροσωπώ τον τομέα των οποροκυπευτικών. Σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τις αγροτικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές για να μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ μετά το 2013. Μα ε, βρίσκομαι και με εκπροσώπους, άλλους εκπροσώπους των του τομέα των οποροκυπευτικών. Μιλήσαμε για την υποστήριξη των οργανώσεων παραγωγών και δόθη το παράδειγμα του τομέα των οποροκυπευτικών παρατηρήσαμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Επίσης, αναλύσαμε τις προτάσεις για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Θα θέλαμε να αναφερθούμε στις αρχές της ΚΑΠ, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές, τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των ε, Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Οργανώσεων και το γεγονός ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα. Επίσης μας ενδιαφέρει το σωστό εισόδημα των γεωργών. Η αγορά των ε, οποροκυπευτικών είναι μία πρότυπη αγορά η οποία θα μπορούσε να παραδειγματίσει και άλλους τομείς παραγωγής. Θα θυμόσαστε ότι στο Πολωνικό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε το γεγονός ότι οι εμπειρίες μας θα χρησιμοποιηθούν σε άλλα τμήματα του τομέα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ο τομέας των οποροκυπευτικών έχει μια καλή διάρθρωση και μέσα στα πλαίσια των συνεταιρισμών, των παραγωγών και των εκμεταλλεύσεων και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τους ίδιους ρυθμούς με τις πιο προηγμένες χώρες. Πρόκειται για μία δυναμική πορεία, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν και θα θέλαμε να βρεθούμε σε μία κατάσταση όπου ο τομέας των οποροκυπευτικών θα είναι τόσο ανταγωνιστικός όσων είναι και σε άλλες χώρες, γιατί πολλές φορές η παραγωγή βρίσκεται σε κατάσταση ανταγωνισμού, κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τις ενδυνάμει αυτές διαδικασίες όμως οι προτάσεις μεταρρύθμισης δεν συνάδουν με αυτά που είπατε κύριε Επίτροπε και σε σχέση με αυτά που είπαν και άλλοι εκπρόσωποι. Η ΚΑΠ και η μεταβατική περίοδος μέχρι ότου τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες δεν εγγυώνται μία σωστή μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς. Θα ήθελα να τα ξανασκεφτείτε όλα αυτά γιατί υπάρχει χρόνος μπορούμε να βρούμε ευεργετικές λύσεις. Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Θα πρέπει να μην επέλθουν αλλαγές πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό θα συνεισφέρει στην καλύτερη ανταγωνιστικότητα του τομέα για να έχουμε καλύτερους όρους εμπορίου για τα οποροκυπευτικά και να βελτιώσουμε και το εισόδημα των γεωργών. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι αναφέρθηκε και το θέμα της διαχείρισης της ε, κρίσης. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα με την κρίση του E. coli και γνωρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικές. Ένα άλλο θέμα είναι οι εξαγωγές. Γνωρίζετε ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν αφορά μόνο την προμήθεια της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να μπορούμε να πολλούμε και προς άλλες αγορές. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλες επιτροπές να ρυθμίσουν ε, μια διαπαντός το θέμα του εμπορίου ως προς τις προμήθειες στη ρωσική αγορά για να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι Τούδε, ο, ε, ένας κύριος που κάθεται στο 115. 115. Κοιτάξτε, στην αρχή εκφράσατε την ικανοποίησή σας γιατί το άζωτο, το κάλιο και τα φωσφατούχα ήταν υπήρξαν υπερβολικής χρήσης. Μπορεί και να συμφωνούσα για τα δύο, αλλά για το κάλιο τα περισσότερα εδάφη στην Ευρώπη δεν έχουν πολύ κάλιο. Δεν πρέπει λοιπόν ως πράσινο μέτρο ή ως μέτρο πρασινίσματος να ζητήσουμε να μειωθεί η περιεκτικό της καλίου στο, στα εδάφη μας. Όσο για τις οργανώσεις των παραγωγών, είπατε να μην καθορίζουν τις τιμές και, να μην υπάρχουν ποσοστώσεις, αλλά φαντάζομαι ότι από δύο πλευρές μπορεί να γίνει επίθεση κατά της πρότασης αυτής. Στο, στη Βρετανία οι οργανώσεις των παραγωγών μερικές φορές μπορεί να γίνουν υπερβολικά μεγάλες οι συνεργατικοί οργανισμοί και αυτό μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες σας προειδοποιώ να το ξέρετε απλώς. Απ' την άλλη αφού λέτε να μην καθορίζουν ποσοστώσεις οι ομαδοποιήσεις παραγωγών. Υπάρχουν τρόφιμα για τα οποία λέμε στους παραγωγούς αν θέλετε να διατηρήσετε τις τιμές να μειώσετε την παραγωγή. Ελπίζω να μην μετρήσετε τέτοιου είδους μέτρα ως ποσοστώσεις διότι το κάναμε με τα αυγά και έτσι σταθεροποιήθηκε η τιμή τους. Πεςτε μας τι φρονείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, Chris Robbins. Chairman. Η κυρία Chris Robbins. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε ε, ε, απογοητευμένη, Δουλεύομαι για τη Life Εκπροσωπώ μια περιβαλλοντική οργάνωση, μία από τις μη κυβερνητικές που αναφέρεται στην ατζέντα σας. Ποιες μη κυβερνητικές θέλετε να ακούσετε. Εάν παίζετε αυτό το παιχνίδι με μας, παίζετε με τα 400 δις ευρώ που υποστηρίζουν αυτή την πολιτική. Μιλάμε για τα χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία υπερασπίζεστε και υπηρετείτε συγκεκριμένα, περιορισμένα συμφέροντα. Όλες οι άλλες ε, μη κυβερνητικέ, δηλαδή το 97% δεν έχει δικαίωμα λόγου. Τι γνώμη έχει ο Επίτροπος γιατί προσπάθησε να εξασφαλίσει το να μπορούν να λάβουν το λόγο όλοι. Τουλάχιστον υπήρχε μία, ένας ανοιχτός διάλογος. Είναι ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός ότι θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπορέσετε να υπερασπιστείτε έτσι μια πολιτική. Δηλαδή μιλάμε για τόσα χρήματα όσα αφορούν τη διάσωση κρατών από τις τράπεζες. Ξέρετε ότι είναι μια πολιτική που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και εμείς θέλουμε να την υπερασπιστούμε παρόλα αυτά. Εμείς ε, τίναμε χείρα ε, βοηθείας, είπαμε ότι θα το υπερασπιστούμε αν υπάρχει ανοιχτός διάλογος και συζητήσαμε πολλά πράγματα και με τους αγρότες. Υπογράψαμε μια κοινή επιστολή με τις αγροτικές οργανώσεις και μια συμβουλευτική επιτροπή Επίσης περιλαμβάνει πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Και τέλος, υπάρχει μια πρόταση επιτάπητος, μια πρόταση πρασινίσματος. Θα θέλουμε κάτι να πούμε ως οργανώσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε το πρασίνισμα. Όλοι λένε φτάνουμε σε δημόσια αγαθά αλλά όχι επαρκή. Γιατί αν δείτε τα στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων, ως προς την κατάσταση της γεωργίας δεν είναι και η χειρότερη δυνατή. Έχουν επέλθει βελτιώσεις, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται ένα δυνατό πρασίνισμα θα πρέπει να εστιαστούμε στο περιβάλλον, όχι στο πάγωμα γεών. Και θα ήθελα να πω στους ευρωβουλευτές, μη σας ε, οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα αυτό το πάγωμα. Δεν είναι το παλαιό πάγωμα, είναι ένα νέο ε, πάγωμα. Μιλάμε για ε, μικρούς υγρότοπους που ήδη υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις σας και δεν θα ήταν ολέθρια αυτά τα αγροτεμάχια για την διατροφική ασφάλεια. Και αυτό δεν φορά μόνο την Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η αγροτική ανάπτυξη, που είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή μόχλευση αυτού του πυλώνα. Εάν δεν έχουμε υποχρεωτικές δαπάνες για τον τομέα του περιβάλλοντος, εάν ε, δεν έχουμε την Natura 2000 της οργανικές καλλιέργειας, δεν θα υπάρξει βελτίωση. Θα ήθελα η Πολωνική Προεδρία που εκπροσωπεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίως και θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Ντεκάστρο και την Επιτροπή Γεωργίας να το λάβουν υπόψη σοβαρά και να μας λάβουν υπόψη διαφορετικά. Επαναλαμβάνετε την παλαιά σας πολιτική και θα προσκρούσετε σε έναν τοίχο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα άλλο μάθημα για το πώς πρέπει να οργανώνουμε τις συζητήσεις όταν μιλάμε για μη κυβερνητικέ και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Όπως ξέρετε, ε, είχε διοναργωνθεί μια τέτοια συνάντηση με τις γερμανικές οργανώσεις. Εάν θέλετε, μπορούμε να συνεργαστούμε και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεχτήκαμε μια σειρά και Εάν λάβετε υπόψη ότι έχουμε δυόμιση ώρες για μια συζήτηση, δεν μπορούμε να ακούσουμε όλες τις οργανώσεις που σχετίζονται με θέματα γεωργίας και αυτό αφορά και τις περιβαλλοντικές. Ε, ο τελευταίος ομιλητής αυτού του τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα είμαι. Για την παραγωγή λυκίσκου που άκουσα ότι αναφέρθηκε προηγουμένως, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι. πρέπει να φροντίσουμε τα επίσημα έγγραφα τα οποία δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως σχετικά ε, με το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν πλέον ενισχύσεις για την παραγωγή λικίσκου. Ως εκπρόσωπος παραγωγών λυκίσκου δεν θα ήθελα να βλέπω τέτοια φαινόμενα. Παρακαλώ λοιπόν βάλτε μια τάξη στο ποια έγγραφα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο γιατί εμείς τις ενισχύσεις τις χρειαζόμαστε για το λυκίσκο. Αυτό είναι το ένα σημείο. Άλλο ένα σημείο που είναι το εξής. Νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετές ευκαιρίες για να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη σε εποχές κρίσης τι θα γίνεται σε μεμονωμένους τομείς. οι διάφορες πολιτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη με κάποιο περιθώριο ευελιξίας το οποίο πρέπει να αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Πήγε εδώ η συζήτηση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει σε μερικά από αυτά που ακούστηκαν. Και όπως γνωρίζετε κύριε Επίτροπε, πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου γενικότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ακόμη μια φορά για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης και για την ευκαιρία που μου δίνεται να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Καταρχήν, χαίρομαι που το θέμα της οργάνωσης, των οργανώσεων των παραγωγών και του ρόλου τους στη διαχείριση των αγορών αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε δεόντως από τους γεωργούς. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους Ισπανούς Αυτά που προτείνουμε είναι κάτι παραπάνω από τα προϋπάρχοντα. Σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα να αναγνωριστούν οργανώσεις παραγωγών διεπαγγελματικά εκτός από τους τομείς που προβλέπονται ρητά από κανονισμούς και που έχουν συγκεκριμένη οργάνωση αγοράς, οπωροκυπευτικά, κρασί και λυκίσκος. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα. Τι σημαίνει αναγνώριση. Ότι αυτόματα θα υπάρχει και εξαίρεση από ορισμένου κανόνες αντιτράστ, δηλαδή το άχθος της αποδείξεως για την ε, θεμητή ή μη λειτουργία της οργάνωσης ως προς τους κανόνες του ανταγωνισμού έχει αντιστραφεί. Δεν πρέπει τώρα οι αγρότες να το αποδεικνύουν. Ο κύριος Άνιο ανέφερε ορισμένες εξαιρέσεις από αυτές τις οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν την παραγωγή τους ανάλογα με τη ζήτηση χωρίς αυτό να θεωρείται παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διοικητικές προκαθορισμένες ποσοστώσεις, αλλά ορισμένες αναγνωρισμένες οργανώσεις μπορούν να σχεδιάσουν την παραγωγή τους ανάλογα με τη ζήτηση, ξαναλέω. Για να κάνουν κοινέ επενδύσεις, να απολύσουν και να διαπραγματευτούν ως οργανώσεις παραγωγών. Ο ρόλος τους λοιπόν ενισχύεται για όλους τους τομείς πια. Αυτό είναι καινούριο. Έπειτα. Μιλήσατε για το έτος αναφοράς και την ανησυχία που νιώθουν οι νέοι αγρότες. Μα το έτος αναφοράς 2011 για τους αγρότες, εκτός από τους καινούριου που εγκαθίστανται τώρα στα χωράφια τους, υπάρχει. Και υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις. Το μόνο που θέλουμε να αποφύγουμε είναι Τώρα που ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει νέος ορισμός των άμεσων πληρωμών γιατί θα συμπεριληφθούν εκεί και νέες γέες, θέλουμε να αποφύγουμε να εμφανιστούν λεγόμενοι αγρότες μόνο και μόνο για να πάρουν τις νέες πληρωμές. Αυτό για το 11 απλώς αλλά φυσικά οι πραγματικοί νέοι γεωργοί που αρχίζουν την ε, δραστηριότητά τους το 2011 θα έχουν δικαίωμα στις πληρωμές αυτές. Για τα ανώτατα όρια, τις οροφές, δώσατε ένα παράδειγμα, όπου όμως δεν τίθεται όπως το είπατε. Όσες οργανώσεις εκπροσωπούν χιλιάδες αγροτών για αυτές υπολογίζεται η πληρωμή ατομικά. Για τις συλλογικές πληρωμές δεν υπάρχει πρόβλημα. Το όριο τίθεται στις ατομικές πληρωμές. Το δικαίωμα. Τώρα για τους λεγόμενους ενεργούς γεωργούς. Και εγώ ήθελα να είναι ο ορισμός πιο συγκεκριμένος αλλά οι προκάτοχοί μου και ολόκληρη η Ένωση είχαν ήδη αναλάβει δεσμεύσει στον ΠΟΕ να μην συνδέσουν τις άμεσες επιχορηγήσεις με την παραγωγή. Το ξέρουν και πολλοί από αυτούς που μίλησαν εδώ. Δεν μπορούμε να βάλουμε στον ορισμό του ενεργού γεωργού κριτήρια που βασίζονται στην παραγωγή ή οποιονδήποτε παράγοντα της παραγωγής δίκτη. Γι' αυτό βάλαμε άλλα στοιχεία για να μπορέσουν να μην συμπεριληφθούν όσοι έχουν γές αλλά δεν τις καλλιεργούν. Κάθε κράτος μέλος προβλέπεται να ορίσει τι είναι η ελάχιστη αναγνωρισμένη δραστηριότητα για να μπορεί ο γεωργός να θεωρηθεί ενεργός. Αυτό έτσι ώστε αν κάποιος γεωργός δεν κάνει τίποτα στη γη του να μην μπορεί να παίρνει και επιχορηγήσεις. Και γιατί βάλαμε ως όριο τα 7.000 ευρώ και όχι κατώτερο. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες, μεσαίες μάλλον εκμεταλλεύσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες και παίρνουν μερικές χιλιάδες ευρώ επιχορηγήσεων γιατί καλλιεργούν ορισμένα εκτάρια αλλά έχουν και άλλα έσοδα. Δεν θελήσαμε αυτούς να τους εξαιρέσουμε από τον ορισμό του ενεργού αγρότη. Τους είπαμε πολυδραστήριους αγρότες. Μερικοί λένε θα χρειαζόταν, θα αρκούσαν 16 σελίδες αντί τόσες πολλές. Αλλά η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύπλοκη. Και βλέπετε και από ό,τι είπαν οι συνάδελφοί σας ότι ο καθένας θέλει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά του και να προστατευτεί. Αν όμως κάπου θέλουμε να είναι κοινή πολιτική, πρέπει οι κανόνες να ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση, αλλιώς δεν είναι κοινή. Γι' αυτό δεν μπορούμε σε 16 σελίδες να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Φιλανδίας ή άλλων χωρών. Η πολυπλοκότητα αυτή βέβαια δεν πρέπει να μας καθιστά τα πράγματα πιο δύσκολα. Όσο δυνατόν περισσότερη απλοποίηση. Το λέει και στην ιστοσελίδα μας. Είναι εκεί ο κατάλογος όλων των στοιχείων απλοποίησης που εφαρμόζουμε. Αλλά το ίδιο αναμένω τώρα να κάνουν και οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ώστε αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσετε επιτόπου να είναι όσο δυνατόν απλούστερα, αλλά να γίνει αυτό από κοινού διότι ακόμη κι αν οι Βρυξέλλες, οι Κομισιόν με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου ορίζουν τους κανονισμούς, η εφαρμογή γίνεται από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Ελπίζω λοιπόν όλοι να κάνουν την ίδια προσπάθεια με την Κομισιόν για να μην γίνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που θα καταθέσουν τροπολογίες. Συμφωνώ ότι μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση αλλά ας μην την κάνουμε ακόμη πιο πολύπλοκη. Για το πρασίνισμα επανέρχομαι γιατί με έκπληξη βλέπω ότι μερικοί εδώ μέσα έχουν ήδη συμμετάσχει σε άλλες συναντήσεις για το θέμα <coughs> όπου αποσαφηνίστηκαν τα πράγματα και ξαναρωτάν τα ίδια για το 7%. Το είπα τρεις φορές ήδη. 7% δεν είναι πάγωμα. Δεν είναι. Ελπίζω να το θυμηθείτε. Ποτέ δεν είπαμε εμείς αυτόν τον όρο. Είπαμε ότι τα 7% είναι για να ληφθούν υπόψη και επιφάνειες γεές που δεν είναι επιλέξιμες αυτή τη στιγμή, που δεν είναι παραγωγικές και που καμιά φορά και οι γεωργοί οι ίδιοι τις εξαιρούν, γιατί είναι ακατάλληλες. Θέλουμε να συνδυάσουμε το στόχο αυτό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, παραγωγής επαρκούς τροφίμων δηλαδή και αύξηση παράλληλα της ανταγωνιστικότητας. Αλλά να μην ξεχνάμε, γιατί ορισμένοι μίλησαν για τη δημόσια συζήτηση που έγινε πέρυσι, κοιτάξτε τι αναμένουμε τι και τι αναμένουν από εμά. Και να γνωρίζετε ότι προτείναμε τον κατάλληλο προϋπολογισμό, αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί σε μια κοινή αγροτική πολιτική που στηρίζει την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα ιδιαίτερα, πρέπει να υπάρχει και σωστή διαχείριση των φυσικών όρων. Θέλουμε να μείνει εθνική δικαιοδοσία η εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων, αλλά αυτό πανενουσιακός. Μπορεί να υπάρχουν πιθανε, δυνατές βελτιώσεις, θα τις συζητήσουμε. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι το 30% που προβλέπετε για το πρασίνισμα είναι μόνο και μόνο για τους γεωργούς, για κανέναν άλλον. Και αυτό το 30% πρέπει να παραμείνει μέσα στις άμεσες πληρωμές των γεωργών. Να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε για να μην εξαιρεθεί. Είναι σημαντικά όλα αυτά και δεν πρέπει να τα λησμονούμε. Αυτά είχα να σας πω και να υπενθυμίσω ότι η πράσινη ανάπτυξη θα διασφαλιστεί με σημαντικά μέτρα, τα οποία είναι μέτρα χωρίς προηγούμενο. Μέτρα τα οποία προβλέψαμε τώρα και συνδέονται με την κοινή αγροτική πολιτική όπου θα συμμετέχει η καινοτομία και θα συνδέεται με την κοινή γεωργική πολιτική. Έτσι θα διασφαλίσουμε την πράσινη ανάπτυξη και βέβαια δεν αποκλείονται οι γεωργικές πρακτικές από αυτό το τομέα γιατί η πράσινη ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από τις γεωργικές πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεκάστρο δεν θέλει να λάβει και πάλι το λόγο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεκάστρο που δεν θέλετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους κυρίες και κύριοι, όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετέσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να ακούσετε τις οργανώσεις αγροτών και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να ακούσετε και είχατε την καλοσύνη και να συνεισφέρετε τις απόψεις σας. Λείπαμε που δεν είχαμε το χρόνο να δώσουμε το λόγο σε όλους και θέλω να ενθαρρύνω τις οργανώσεις των αγροτών να συνεχίσουν αυτή τη συζήτηση και να την κρατήσουν ζωντανή στις περιφέρειές τους, στις χώρες τους, γιατί πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ζητήσετε από τους υπουργούς σας και από τους βουλευτές στη χώρα σας να συμμετέχουν και εκείνοι στη συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, οι αποφάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ θα ληφθούν ισομερώς από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν αυτή η συζήτηση να παραμείνει ζωντανή και πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα επηρεάσετε εσείς το μέλλον της ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie, Marek. Very well indeed. But it's always like this, you know, when you invite 10, you should invite